Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Προτού υποδεχθούμε επισήμως και τον πρόεδρο Μπατιστέλη, ας περάσουμε πρώτα στο σημείο 1, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε κάνει κάποιες μικρές αλλαγές. Το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή η ανταλλαγή απόψεων για την αίτηση άρσης της κομβελτικής ασυλίας του Ντανίκα έχει ακυρωθεί μετά από αίτημα του ίδιου του εισηγητή. Το σημείο 16, πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας νομοθεσίας REFIT, τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές, με εισηγήτρια την κυρία Κάουφ Αφμαν, θα καλυφθεί στο τέλος, μετά τις ψηφοφορίες δηλαδή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσει, εναλλακτικέ προτάσει για αυτέ τι αλλαγέ. Αν όχι, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Δεν υπάρχουν περαιτέρω ανακοινώσει του Προέδρου. Uh, we should also uh, approve our minutes Πρέπει να εγκρίνουμε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16ης Απριλίου, καθώς επίσης και τη συνεδρίαση της 6ης και 7ης Μαΐου. Υπάρχουν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις. Δεν βλέπω κανέναν, συνεπώς εγκρίνουν τα πρακτικά. Μπορούμε συνεπώς να περάσουμε στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία, τον κύριο Μπενουά Μπατιστέλη. Όπως ξέρετε, πρόσφατα μία αντιπροσωπεία της επιτροπή μας πήγε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία, Μας υποδέχθηκε εκεί ο πρόεδρος Μπενουά Μπατιστελή και νομίζω ότι και η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Μπατιστέλη στη δική μας την Επιτροπή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, δεδομένη της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία ακύρωσε την προσφυγία ακύρωσης κατά της ενισχυμένης συνεργασίας όσον αφορά το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Κύριε Μπατιστέλη, κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και σας δίνω αυτής αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τη δυνατότητα να βρίσκομαι σήμερα στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον Πρόεδρο Σβόμποντα που μου δίνει την εξαιρετική αυτή ευκαιρία να σας ενημερώσω για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθώς επίσης και για τις προτεραιότητές μας και για τους στόχους μας. Ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία. Από τότε που εξελέγει ενό πρόεδρο του EPO είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σα. Και συνεπώ θα ήθελα να σα πω ότι η δική σα Επιτροπή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, έχει διδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στην όλη διαδικασία που οδήγησε στην ε, υλοποίηση του ενιαίου δίπλωμα ευρεσιτεχνία καθώ επίση και στι σχετικού κανονισμού η ε, δέσμη μέτρων για το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για την Ευρώπη. Θα προωθήσει την κοινοτομία στην Ευρώπη και την καταστήσει πιο ανταγωνιστική σε σχέση με την Ασία και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τι νέε προκλήσει που αποκύπτουν από την δέσμη αυτή μέτρων όσον αφορά το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία και κατά αυτόν τον τρόπο θα ανταποκριθούμε σε όλε τι υποχρεώσει μα και σε όλε τι νέε αρμοδιότητε που προκύπτουν. Θα ήθελα λοιπόν να αφαιρθώ καταρχά στο έργο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία και στη συνέχεια να αναφερθώ στι τελευταίε εξελίξει που είχαμε όσον αφορά το ενιαίο σύστημα διπλώματο ευρεσιτεχνία και στη συνέχεια θα αναφερθώ επίση και στην περαιτέρω εναρμόνιση που προβλέπεται στα πλαίσια του ενιαίου διπλώματο ευρεσιτεχνία. Το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι ουσιαστικά μία απλή σύμβαση ανάμεσα στην κοινωνία και τους εφευρέτες. Το σύστημα λοιπόν αυτό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας βασίζεται σε μια βασική οικονομική συναλλαγή, ένα κοινωνικού οικονομικού συμβολέου ανάμεσα στους εφευρέτες και την κοινωνία. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δίνει στον κάτοχό του ένα προσωρινό δικαίωμα να αποκλείσει κάποιους άλλους ανθρώπους από να χρησιμοποιούν την εφεύρεσή του. Η αποκλειστικότητα αυτή δημιουργεί λοιπόν μια πλεονεκτική θέση στην αγορά για αυτόν τον κάτοχο διπλώματο ευρεσιτεχνία και του δίνει τη δυνατότητα να έχει τα απαραίτητα κίνητρα για να δημιουργήσει μια εφεύρεση η οποία θα είναι σημαντική για την οικονομία και την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο κάθε εφευρέτης να περιγράφει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια την εφεύρεσή του και στη συνέχεια από τη στιγμή που πέσουν στο δημόσιο τομέα πληροφορίες αυτές μπορεί οποιοδήποτε μελλοντικό εφευρέτης να βασιστεί στις πληροφορίες αυτές για να δημιουργήσει τη δική του εφεύρεση, μια περαιτέρω εξέλιξη στην τεχνολογία. Ξέρετε ότι πολύ συχνά οι εφευρέτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την εναλλακτική νομοθεσία του εμπορικού απορρίτου. Εσεί ξέρετε ότι επεξεργάζεστε μια σχετική πρόταση. Τα πράγματα όμως είναι εξίσου πολύπλοκα, σημαίνει ότι πρέπει κανείς να διαρθρώσει την εργασία στα πλαίσια της επιχείρησής του, αλλά και στα πλαίσια της σχέσης που έχει με πελάτες και υπεργολάβους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει καμία διαρροή πληροφορίας. Και εφόσον χρησιμοποιείτε παράλληλα ένα άλλο σύστημα διατήρησης πληροφοριών, ενδεχομένως να μην μπορείτε να έχετε ένα απόλυτο σύστημα προστασίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει το απαραίτητο ε, πλαίσιο προστασίας το οποίο παρέχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Τα διπλώματα ευρεστεχνίας όμω ωφελούν και την ίδια την κοινωνία όσον αφορά το ζήτημα τη καινοτομία, του ανταγωνισμού, τη οικονομική ανάπτυξη και τη κοινωνική πρόνοια. Όσον αφορά το κοινωνικό αυτό συμβόλαιο ενό διπλώματο ευρεστεχνία, ουσιαστικά η κοινωνία παραχωρεί προς τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας την αποκλειστική την αποκλειστικότητα, ένα αποκλειστικό δικαίωμα για να χρησιμοποιεί την εφεύρεσή του αυτή, προκειμένου να δημιουργηθούν τα απαραίτητα κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω καινοτομία, αυτό είναι αρκετά θετικό γιατί κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η επιλογή των καταναλωτών, αυξάνεται η οικονομική ανάπτυξη καθώς επίσης και η κοινωνική πρόνοια. Δημιουργείται επίσης οικονομική μεγένθηση, νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση έχουμε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Επίσης έχουμε μια διάχυση όλων των απαραίτητων τεχνολογικών πληροφοριών που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω εφευρέσεις. Προκειμένου να κάνει κανείς αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει ο Εφευρέτη να υποβάλει μια πλήρη αίτηση με πλήρη περιγραφή της εφεύρεσης αυτής. Ε, οι υπόλοιποι πολίτες μπορούν να αποφεληθούν από τις ε, γνώσεις αυτές και να δημιουργήσουν και αυτοί με τη σειρά τους νέες εφευρέσεις. Το ονομάζουμε αυτό σορευτική γνώση. Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε αυτό που είχε πει ο Ισαάκ Νιούτον, ότι βασιζόμαστε, στεκόμαστε ως είναι πάνω στους ώμους των γιγάντων και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εφεύρουμε περισσότερο. Πρέπει όμως να δούμε επίση και ποιε είναι οι οικονομικέ επιπτώσει όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σε συνεργασία με το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς το Σεπτέμβριο του 2013 κοινοποιήσαμε μία δημοσιοποιήσαμε συγχωρείτε μια κοινή μελέτη προκειμένου να φερθούμε σε αυτές τις, στους βιομηχανικούς κλάδους που χρησιμοποιούν πολλά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναλύσαμε πολλούς διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς και προσπαθήσαμε συγκρίνοντα βάσει δεδομένων, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι επαγγελματικοί κλάδοι που χρησιμοποιούν περισσότερο εμπορικά σήματα, μοντέλα, πρότυπα, καθώς επίσης και άλλες μορφές ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα κάποια αριθμητικά δεδομένα, ιδίω ε, όσον αφορά κάποιους μακροοικονομικούς ε, δείκτες. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι περίπου ένα 40% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργείται από τους κλάδους αυτούς που χρησιμοποιούν εντόνως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αντιστοιχούν επίσης αυτοί οι φορείς, αυτοί οι επαγγελματικοί κλάδοι σε ένα 35% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποίησαμε και κάποιους άλλους δείκτες και πάντως για πρώτη φορά καταφέραμε να ποσοτικοποιήσουμε τον οικονομικό αντίκτυπο από μακροοικονομικής πλευράς όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ας αναφερθούμε τώρα πιο συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Ποιοι είμαστε και τι ακριβώς κάνουμε. Αποστολή μας είναι να κατοχυρώσουμε διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να διαχέουμε τις ε, σχετικές πληροφορίες και μέσω της δραστηριότητας αυτής, της δυτής αυτής δραστηριότητας, καταφέρνουμε να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα, την κοινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη παντού στην Ευρώπη, μέσω μιας δέσμευσής μας για αποτελεσματικές και υψηλά ποιοτικές υπηρεσίες. Βλέπετε εδώ πέρα στο χάρτη αυτό τις χώρες τις οποίες δραστηριοποιούμεθα. Δεν είμαστε οργανισμός του Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε ένας διακυβερνητικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από μια συνθήκη που υπογράφει το 1973 το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρωστεχνίας άρχισε να εργάζεται το 1978. Τότε ήμασταν μόνο 7 χώρες, τώρα είμαστε πλέον 38 χώρες και συμμετέχουν, μάλλον πρόκειται να, αρχίσουν να, προσχω... να... να προσχωρήσουν δύο χώρες, το Μαυροβούνιο και η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και πρόσφατα υπογράψαμε μία συμφωνία με το Μαρόκο, σύμφωνα με την οποία το Μαρόκο από την 1η Μαρτίου του 2015 αρχίζει και αναγνωρίζει και αυτό ως εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Και νομίζω πραγματικά ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αυξήσουμε την γεωγραφική μας επιρροή χωρίς από την άλλη να θέτουμε κάποιο όριο όσον αφορά τον αριθμό των κρατών μελών που θα μπορούσαν να προσχωρήσουν. Είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη διακυβερνητική οργάνωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 7.000 άτομα εργάζονται για μας, εκ των οποίων τα 4.250 είναι ε, υψηλά εξειδικευμένοι μηχανικοί και επιστήμονες, είναι οι λεγόμενοι ελεγκτές, οι εξεταστές, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι επεξεργάζονται όλες αυτές τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τις οποίες λαμβάνουμε. Είμαστε ένας αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός, πράγμα το οποίο σημαίνει δεν λαμβάνουμε καμία χρηματοδότηση ούτε από τα κράτη-μέλη, αλλά ούτε και από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό, και όχι μόνο τον εξαρτώμεθα χρηματικά από τα κράτη-μέλη, αλλά παράλληλα εμείς καταφέρνουμε και δημιουργούμε τους δικούς μας πόρους, καθότι μοιραζόμαστε τελικά με τα κράτη-μέλη το ίμιση των τελών, τα οποία προκύπτουν από τα διπλώματα βρεστεχνίας. Από αυτόν τον ετήσιο προπολογισμό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, 400 εκατομμύρια ευρώ τελικά επιστρέφουν στα κράτη-μέλη με τη μορφή εσόδων. Είναι χρήματα τα οποία πηγαίνουν από το δικό μας το γραφείο προς τα κράτη-μέλη. Βλέπετε εδώ πέρα τα βασικότερα σημεία όσον αφορά τη δραστηριότητά μας, όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Βλέπουμε ότι είναι μια τάση η οποία παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια. Στην αυξητική αυτή τάση συμμετέχει προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπετε ότι κατά μέσο όρο έχουμε αυξήσει τα τελευταία 15-20 χρόνια κατά 3,1% τον αριθμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τα οποία φτάνουν σε εμά. Έχουμε φτάσει τις 274.174 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Από πού προέρχονται όλες αυτές οι αιτήσει. Βλέπετε εδώ πέρα ένα γράφημα το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το 65% των αιτήσεων αυτών έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα 35% προέρχεται από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης για να είμαι πιο ακριβή. Βλέπετε εδώ πέρα ότι οι περισσότερες αιτήσει φτάνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η τέταρτη κατά σειρά χώρα όσον αφορά τις αιτήσει. Ακολουθεί η Ιαπωνία, στη συνέχεια η Γερμανία, η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην κατάταξη αυτή με 11%. Στη συνέχεια έχουμε την Κίνα με 9%, την Κορέα με 6% και τη Γαλλία, τη δεύτερη δηλαδή μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης με 5%. Για ποιο λόγο βλέπουμε όλες αυτές τις αλλαγές, όλες αυτές τις εξελίξεις. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πριν από τρία χρόνια η Κίνα βρισκόταν στο επίπεδο της Γαλλίας, δηλαδή με ένα 5% του συνόλου των αιτήσεων διπλωμάτων της και μέσα σε τρία μόνο χρόνια κατάφερε να αυξήσει τις αιτήσει της κατά 80% η Κίνα, ενώ η Γαλλία σταθεροποίησε τελικά την θέση την οποία κατήχε. Ποια είναι η στρατηγική που ακολουθούμε τώρα στο δεδομένο αυτό περιβάλλον. Προτεραιότητά μα είναι να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε την υψηλή ποιότητα των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Όταν λέμε ποιότητα, αυτό που εννοούμε είναι διπλώματα ευρεσιτεχνία τα οποία θα έχουν μια σωστή νομική βάση, τα οποία από νομική πλευρά θα στέκουν. Δεν μα ενδιαφέρει τόσο πολύ η εμπορική, η οικονομική πτυχή των διπλωμάτων αυτών ευρεσιτεχνία, αυτό είναι περισσότερο αρμοδιότητα των ίδιων των επιχειρηματιών. Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιούμε ένα μέσο, ένα εργαλείο το οποίο θα είναι νομικά ισχυρό και θα αποτελεί πραγματικά προστιθέμενη αξία για τη στρατηγική τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ποιότητα μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να κάνει τελικά τη διαφορά και να καταστήσει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οικονομικά βιώσιμο. Η στρατηγική μας βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, επικεντρωνόμαστε όπως σας είπα στην ποιότητα, Επιθυμούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας και επιθυμούμε επίσης να συμβάλλουμε όλο και περισσότερο σε μια εναρμόνιση του παγκόσμιου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Γι' αυτό το λόγο εγκρίναμε πέντε οδικούς χάρτες με την υποστήριξη των 38 κρατών μελών που συμμετέχουν στο EPO. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο η δική μας παραγωγικότητα και κάθε φορά βέβαια που υπάρχουν και αλλαγές Υπάρχουν προφανώς και κάποιες αντιρρήσεις ή αμφιβολίες. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν συμφωνούν με τις εξελίξεις αυτές. Αλλά αυτό αποτελούσε ανέκαθεν χαρακτηριστικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία. Πολλές φορές βέβαια αντιρρήσεις αυτές έφτασαν στα άκρα και πολλές φορές έθεσαν να αμφιβόλο την αποτελεσματικότητα της εργασίας του ΕΠΟ. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα εργασίας του EPO είναι απόλυτα διαφανές, όλες μας οι δράσεις παρουσιάζονται με τον πιο λεπτομερή τρόπο και έχουν εγκριθεί και έχουν υποστηριχθεί από τα κράτη-μέλη μας. Έχουμε δηλαδή μια ομόφωνη υποστήριξη από τα 38 κράτη-μέλη όσον αφορά αυτόν τον οδικό χάρτη που παρουσιάσαμε τον Ιούνιο του 2014. Επίσης, οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί για λίγους μονομήνες και παρόλα αυτά οδήγησαν σε πολύ απτά θετικά αποτελέσματα για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Οι μεταρρυθμίσεις μας επίσης βασίζονται στις κοινά αποδεκτές βασικές αρχές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθήσαμε προφανώς την νομολογία της δικαστικής μας αρχής που είναι το Διοικητικό Δικαστήριο του ε, Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Σας υπενθύμισα λοιπόν εν συντόμω τη στρατηγική μας, να σας δώσω τώρα και κάποια παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα που θα ήθελα να σας δώσω αφορά μια νέα υπηρεσία που λέγεται μετάφραση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουμε εισαγάγει πρόσφατα. Ε, τώρα, ε, για να σας παρουσιάσω λίγο τη σημασία αυτού του νέου εργαλείου, θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό το οποίο καθορίζει την ποιότητα ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι ε, πόσο πλήρης έρευνη έχει γίνει επί της αιτήσεως ε, για να είμαστε βέβαιοι ότι η συγκεκριμένη εφεύρεση είναι πραγματικά κάτι νέο. Ε, αυτό το αποκαλούμε κριτήριο καινοτομία. Και φυσικά αυτή η έρευνα θα πρέπει να γίνει όχι μόνο μέσω προηγούμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αλλά ε, παντού. Αυτό το αποκαλούμε στις διαθέσιμες γνώσεις μας. Και ε, δεδομένου ότι έχουμε όλο ένα και περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνία τα οποία έχουν συνταχθεί σε ε, μη ευρωπαϊκέ γλώσσε, μία από τις βασικές προκλήσεις είναι αυτό το εμπόδιο της γλώσσας. Ε, υπάρχουν περισσότερα κοινόζικα διπλώματα ευρεσιτεχνία, ιαπωνικά διπλώματα ευρεσιτεχνία και επομένω είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτύχουμε το σκοπό μα. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέπουν όχι μόνο ε, σε εμά ως ε, άνθρωποι που εξετάζουν τα ε, διπλώματα ευρεσιτεχνία, αλλά και σε όλη την επιστημονική κοινότητα να έχει πρόσβαση σε αυτές τις διαθέσιμες γνώσεις. Γι' αυτό ακριβώ και έχουμε αναπτύξει μια νέα υπηρεσία που λέγεται Patent Translate σε συνεργασία με την Google και είμαστε το μόνο γραφείο ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παγκοσμίω, το οποίο παρέχει στην ιστοσελίδα του δωρεάν 24 ώρες 24 ώρες τέτοιες υπηρεσίες. Καλύπτει 32 γλώσσες, 28 γλώσσες κρατών μελών, καθώς επίσης και τις τέσσερις μεγάλες γλώσσες ε, στην επιστήμη και στην τεχνολογία, κινέζικα, ιαπωνικά, κορεατικά και ρώσικα. Η υπηρεσία αυτή δεν χρησιμοποιείται μόνο από τους εξεταστές μας και από τα άλλα ε, γραφεία και τους άλλους εξεταστές, αλλά χρησιμοποιείται και από το ευρύτερο κοινό. Έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής και έχουμε πλέον 23.000 ε, αιτήματα ε, μετάφρασης ημερησίως. Βεβαίως αυτό Αυτές οι μεταφράσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ, αλλά μας επιτρέπουν να αναζητήσουμε τα σχετικά έγγραφα σε αυτό το τεράστιο όγκο ε, εκατομμυρίων σελίδων και από εκεί και πέρα, εάν κάποιος ε, θέλει να προσδώσει νομική αξία στα στοιχεία αυτά, ε, τότε θα πρέπει να λάβει μια επίσημη μετάφραση από ειδικού μεταφραστέ. Ένα άλλο παράδειγμα στοιχείων που αναπτύσσουμε ε, με φέρνει σε αυτή την ενία ε, το νέο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρωστεχνίας. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν ε, συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρωστεχνίας πριν από 20 χρόνια, ήμασταν σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Τότε δημιουργήθηκε ένα σύστημα με μια κεντρική αρχή, το οποίο παρήχε ένα ενιαίο δίπλωμα ευρυστεχνίας, το οποίο ίσχυε για όλα τα κράτη-μέλη. Η ισχύ αυτή όμω δεν προσδίδεται αυτόματα. Όταν κάποιο κατέχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνία, θα πρέπει να αποφασίσει σε ποια χάρη, ε, χώρα συγγνώμη, θα θέλει να επικαιρώσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνία του. Και από εκεί και πέρα η όλη διαδικασία επικύρωση ε, μετατρέπει το ευρωπαϊκό δίπλωμα Ευρυστεχνία είναι ένα εθνικό δίπλωμα Ευρυστεχνία. Αν επικυρώσετε για παράδειγμα ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα Ευρυστεχνία στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στι κάτι χώρε που είναι οι τέσσερι χώρε οι οποίε επικυρώνουν τα περισσότερα διπλώματα Ευρυστεχνία, το δίπλωμα ευρυστεχνία σα γίνεται και ένα γερμανικό, γαλλικό, αγγλικό και ολλανδικό δίπλωμα Ευρυστεχνία. Και από εκεί και πέρα υπόκειται στα εθνικά δικαστήρια σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές. Και βέβαια τα δικαστήρια μπορεί να λάβουν διαφορετικές αποφάσεις. Επομένως, εν τέλει, ξεκινώντας από ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, έχετε διαφορετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ήδη λοιπόν, στη δεκαετία του 70, είχαμε προβλέψει να συμπληρωθεί αυτό το πρώτο τμήμα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρωσιτεχνίας, όπως το γνωρίζουμε εδώ και 40 περίπου χρόνια, μέσω ενός τεράστιου βήματος που σήμαινε ότι θα έχουμε ενωσιακό ε, δίπλωμα ευρωσιτεχνίας. Και αυτό αποφασίστηκε μετά από δεκαετίες συζητήσεων, μέσω αυτού του προγράμματος ενισχυμένης συνεργασίας και της έγκρισης των ευρωπαϊκών κανονισμών που δημιουργούν αυτό το ενωσιακό δίπλωμα ευρυστεχνίας. Και αυτό συνδέεται και με μια συμφωνία για να δημιουργήσουμε το νέο ε, ενοποιημένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να υπάρχει και ένα ε, ενοποιημένο δικαστήριο. Ε, ποιος είναι ο βασικός στόχος λοιπόν και κατά πόσον επιτεύχθη αυτός από το ενωσιακό διαβατήριο. Αυτός έχει επιτευχθεί διότι θα είναι ένα ευρω... Ε, ενωσιακό διαβατήριο το οποίο θα χορηγείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλώματος της και θα θεωρείται επικυρωμένο μέσω μιας τυπικής διαδικασίας ε, του Ευρωπαϊκού ε, Γραφείου Διπλωμάτων Ευρωσιτεχνίας και θα ισχύει και στις 25 χώρες μέλη που συμμετέχουν. Ένα βασικό στοιχείο το οποίο συμβάλλει στην επιτυχία του Διπλώματος Ευρωσιτεχνίας είναι ότι προσφέρουμε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιλογή μεταξύ διαφόρων μορφών προστασίας. Μπορεί να επιλέξουν εθνική προστασία, την κλασική ευρωπαϊκή προστασία και επίσης μπορούν να επιλέξουν και μια τρίτη λύση που είναι ε, ε, προστασία ενωσιακού ε, διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Προαδέχεται λοιπόν αυτή η ευελιξία ώστε να επιλέξουν το εργαλείο το οποίο είναι το πλέον κατάλληλο με βάση τη στρατηγική τους. Και αυτό το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποτελεί πολύ μεγάλη απλούστευση σε σχέση με το τρέχον σύστημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, διότι υπάρχει μόνο ένα διοικητικό ε, βήμα το οποίο θα πρέπει να γίνει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλώματος Εργασίας για να υπάρχει ε, προστασία σε 25 χώρες αντί να πρέπει να γίνουν 25 εθνικές διαδικασίες διατυπώσεων. Και αυτό φυσικά ε, σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μείωση στο κόστος και φυσικά θα είστε και σε θέση να καθορίσετε και τα τέλη ε, κατά τρόπον ώστε εάν τα δούμε μπορούμε να είμαστε σε μία μείωση της τάξης του 70% σε σχέση με την παρούσα κατάσταση. Τέλος, θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου, διότι αντί να υπάρχουν τελείως διαφορετικές ε, νομολογίες θα υπάρχει ένα ενιαίο δικαστήριο το οποίο κάθε χρόνο θα δημιουργήσει την νομολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα είναι η ίδια για όλους τους ε, ε, ενδιαφερομένους. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο θα συμπεριληφθεί στο σύστημα μέσω της εφαρμογής ε, αυτού της νέας προστασίας του ενωσιακού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Πού βρισκόμαστε τώρα λοιπόν, τρία χρόνια μετά τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει υπάρξει καλή πρόοδος όσον αφορά το λεγόμενο UPC, το ε, δικαστήριο λοιπόν ε, για τα ε, ενωσιακά διπλώματα ευρεσιτεχνίες. θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή μια διαδικασία επικύρωσης. Χρειάζονται 13 κυρώσει από τις 25 ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή και να ξεκινήσει τη λειτουργία του το δικαστήριο. Μέχρι τώρα έχουμε κύρωση από 7 χώρες, συμπεριλαμβάνεται και η Γαλλία. Χρειαζόμαστε 13 ε, που θα περιλαμβάνουν και τις τρεις μεγαλύτερες χώρες, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι με την απόφαση που ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον περασμένο μήνα, το οποία όπως επεσήμανε και ο πρόεδρός σας ε, ε, στην εισαγωγή αυτής της συζήτησης, θεωρούμε πολύ σημαντική, διότι διευκρινίστηκε το τελευταίο νομικό πρόσκομα και διασκεδάστηκαν οι ανησυχίες ώστε να καθοριστεί ότι η νομική βάση του συστήματος αυτού είναι η σωστή, συμμορφούται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και επομένως μπορεί πλέον να εφαρμοστεί χωρίς ε, να υπάρχει κάποιος νομικός κίνδυνος. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αποτελέσει την κατάλληλη όθεση ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των χειρώσεων και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε και χορήγηση του πρώτου ενωσιακού διπλώματος ευρωτεχνίας ήδη από το χρόνο, από το 2016. Υπάρχει ένα ακόμα σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί και αφορά το ίδιο το ενωσιακό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το ύψος των τελών, ώστε να καθορίσουμε και τι θα γίνεται με το ετήσιο τέλος που πρέπει να καταβάλλεται αυτή στιγμή χορηγηθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εάν κάποιος δεν πληρώσει το ετήσιο τέλος, χάνεται το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και πλέον γίνεται δημόσιο, ε, δημόσια εφεύρεση. Αντί λοιπόν να έχουμε καταβολή 25 εθνικών αιτήσεων τελών, όπως γίνεται τώρα, Λοιπόν, δεν χρειάζεται πλέον να έχουμε 25 διαφορετικά τέλη και δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να τα προσθέσουμε, θα πρέπει να καθοριστεί ένα επίπεδο τελών, το οποίο ε, θα είναι και δέλεαρ για τις επιχειρήσεις. Μετά από αρκετές συζητήσεις και πολλές προσωμιώσεις, ε, η απόφαση θα ληφθεί από τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή Select, που είναι ένας φορέας ε, που είναι τμήμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και τους προτείνουμε να καθοριστούν αυτά τα τέλη ε, στο επίπεδο των λεγόμενων ε, μεγαλύτερων τεσσάρων, που σημαίνει ότι θα προσθέσουμε τα τέλη των τεσσάρων χωρών που έχουν τις περισσότερες επικυρώσεις, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις κάτω χώρες, και για το κόστος αυτών των τεσσάρων θα παρέχεται προστασία σε 25 χώρες. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι θα χρειαστεί σίγουρα και υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι η πρώτη προτεραιότητα για αυτό το ενιαίο δίπλωμα ευρυστεχνίας δεν είναι να υπάρχει ε, συνένεση για τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνία, αλλά να είναι κατάλληλο και να υπάρχουν έσοδα για τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνία, αλλά να υπάρχει κάποιο δέλεαρ για τι επιχειρήσει, επομένω να έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερα τέλη ε, για να μπορέσουν να υποβάλουν και αρκετέ επιχειρήσει ε, αιτήσει για διπλώματα ευρεσιτεχνία. Αυτό θα αποφασιστεί μέχρι το τέλος του μήνα, γεγονός το οποίο θα μας επιτρέψει να ε, δώσουμε και το πρώτο ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 2016 όταν θα ξεκινήσει και η λειτουργία του συστήματος. Τώρα θα ήθελα να ολοκληρώσω με τις ε, πολυμερείς προκλήσεις που έχουμε. Εδώ έχουμε διάφορα κριτήρια για την λήψη διπλώματο ευρεσιτεχνία και του βασικού κανόνε ε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Για παράδειγμα, οι κανόνε είναι αρκετά διαφορετικοί στι ΗΠΑ από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε λοιπόν να ενερμονίσουμε αυτού του κανόνε και τι διαδικασίε και τι διάφορε πρακτικέ, ώστε να πλουστεύσουμε τη ζωή των χρηστών, των επιχειρήσεων και να τους επιτρέψουμε να χρησιμοποιούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τους σε όλο τον κόσμο. Η εναρμόνιση βέβαια είναι μια μακρά διαδικασία, δεν μπορεί να γίνει εν μία ανοιχτή και εργαζόμαστε σε διάφορα επίπεδα ώστε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία εναρμόνισης. Το ένα επίπεδο είναι περισσότερο τεχνικού και διαδικαστικού χαρακτήρα. Έχουμε συστήσει ε, μια άτυπη ομάδα, την IP5, η οποία περιλαμβάνει τα πέντε μεγαλύτερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ε, τι Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Κορέα και την Ευρώπη. Και εδώ ε, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίων αποτελεί τη φωνή της Ευρώπης και έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε λίγο και τις εξελίξεις του παγκόσμιου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά το σύστημα και υπάρχει πρόοδος. Για παράδειγμα, ε, θα συσταθεί το, η λεγόμενη παγκόσμια υποβολή φακέλου. Δηλαδή, με ένα φάκελο θα μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση σε ε, διάφορα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Υπάρχουν ε, και κάποιες άλλες τεχνικές πρόοδοι, αλλά δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις για αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο. Υπάρχει και μία ακόμα διάσταση εναρμόνισης ε, η εναρμόνιση για το ουσιαστικό δίκαιο που αφορά τους κανόνες και τις αρχές, ε, στοιχείο που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν είναι άμεση αρμοδιότητα του γραφείου και ούτε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει μία πρόκληση να επιλέξουμε κατά πόσο θα γίνουν διμερείς συζητήσει, για παράδειγμα με τις ΗΠΑ, ή αν θα πρέπει να ευνοήσουμε πολυμερείς λύσεις. Και το θέμα αυτό το έχουμε συνδυάσει και με τις διαπραγματεύσεις για την TTIP, οι οποίες είναι εξελίξη. Ξέρω ότι η Επιτροπή σας και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά τις συζητήσεις για την TTIP και θεωρώ ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικά θετικό και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για το ενδιαφέρον σας. Το ενδιαφέρον που εκφράζεται για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά το θέμα των ε, πνευματικών δικαιωμάτων, δεν θεωρούμε ότι ε, ιδίω για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία, η TTIP είναι καλό μέσο για να υπάρξει εναρμόνιση. Δείτε επίσης και τι ενδιαφέρον υπάρχει από τους Ευρωπαίους ε, ε, για την ε, πρόοδο αυτής της εναρμόνισης. Υπάρχει ένα φόρουμ το οποίο επιτυγχάνει κάποια πρόοδο, αν και αργή πρόοδο, είναι η ομάδα της WIPO, που είναι ένας διεθνής οργανισμός διπλωμάτων τεχνίας, παρακλάδι της οικογένειας των Ηνωμένων Εθνών και ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα είναι μια υποδομάδα ε, την οποία αποκαλούμε B+, και εκεί υπάρχει κάποια πρόοδο στα θέματα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω λοιπόν με αυτή την παρουσίαση, τονίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχημένη ιστορία. Τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο ε, βοήθησε την καινοτομία, γεγονός το οποίο έφερε την Ευρώπη στα ενία της ε, διαδικασίας ε, χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παγκοσμίω. Θα κορυφωθεί λοιπόν αυτή η δράση με αυτό το ενωσιακό δίπλωμα Ευρεσιτεχνία και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία είναι περήφανο διότι του ανατέθηκε η χορήγηση και η διαχείριση αυτού του πολύ σημαντικού εργαλείου για την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή οικονομία και ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει τη. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την προσοχή σα και ε, με τα χαρά να απαντήσω και στι ερωτήσει σα ή να ακούσω τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίασή σας που ήταν πάρα πολύ επικοδομητική θα έλεγα για τους ευρωβουλευτές μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Μπορείτε να βασίζεστε και ομιλώ εξ ονόματος των μελών αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στην υποστήριξή μας όσον αφορά το θέμα των τέλων και το να πιστούν τα κράτη-μέλη όσον αφορά αυτό το εγχείρημα και σας ευχαριστούμε και πάλι. Και τώρα, χωρίς να καθυστερούμε, ερωτώ τους ευρωβουλευτές μας. Έχουν κάποιες ερωτήσεις ή αιτήματα κάποιος να παρέμβει. Ο Αξερφός παρακαλώ. Λειτουργεί έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά για την εισήγησή σας. Περιμένω μια στιγμή να φορέσετε τα ακουστικά σας. <laughs> Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την εισήγησή σας. Νομίζω μας καθιστά σαφές πόσο σημαντικό είναι το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών για την οικονομία μας. Και είναι πολύ καλό το ότι μας τα εξηγήσατε αυτά. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο φυσικά είναι <clears throat> τα προβλήματα τα οποία αναφύονται και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αφενός το αναφέρατε, το TTIP. Φαίνεται ότι σωστά συνετά αντιδράσαμε από πλευράς ε, Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνοδευτικά, αλλά για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν φαίνεται ότι εφαρμόζονται τα πράγματα όπως θα, θα επιθυμούσαμε και σε σχέση με τις φιλοδοξίες μας. Δεν γνωρίζω αν τα κράτη-μέλη τώρα έχουν μια βραδύτερη διαδικασία επικύρωσης ή αν θα υπάρχει, δεν, αναγνωρίζουν μήπως το προτέρημα, τα προτερήματα ενός ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αυτό το οποίο με παραξενεύει είναι η αντιπαράθεση για τα τέλη αλλά εγώ θα έλεγα προσωπικά ότι δίνει κάποιο προτέρημα αυτό το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Παίρνουμε τα τέλη από τα πρώτα τέσσερα κράτη που έχουν τα περισσότερα διπλώματα. Καλύπτονται όμως και τα 25 κράτη και έτσι είναι ένας πολύ καλός συμβιβασμός αν μπορεί κανείς να πει ότι εντάξει ωραία θα μπορέσουμε με τα κόστη να ε, βρούμε μια λύση και αυτό θα μας δώσει και οικονομικά προτερήματα. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, οι επιχειρήσεις ή εκείνοι που το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ε, το καταθέτουν δεν θα είναι πρόθυμοι να επιλέξουν ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αν τα τέλη είναι υπερβολικά υψηλά. Γι' αυτό θα έλεγα εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο φυσικά θα έπρεπε να πιέσουμε να προαθεί το ενιαίο δίπλωμα βρεσιτεχνίας και να καταστήσουμε σαφές ότι εδώ δεν μπορεί να αποτύχει το εγχείρημα λόγω των τελών, αν θα έχουμε δηλαδή ένα ενιαίο δίπλωμα βρεσιτεχνίας ή όχι. Πρέπει για τα οικονομικά συμφέροντα αυτό να είναι επικερδές και υποφελές για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό αυτή η πρόταση για την οποία έγινε λόγος, <clears throat> δηλαδή για τα τέσσερα στους τέσσερις ε, ε, μεγαλύτερους ε, που θα συμμετέχουν είναι ένα επιχείρημα και θα έπρεπε να ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών με ταχύς ρυθμούς να υλοποιήσουν την πρόταση αυτή, γιατί είναι μια θετική ισορροπία μεταξύ των οικονομικών συμφερόντων και των νομικών προσεγγίσεων. Και δεν πρόκειται για τα ξεχωριστά συμφέροντα των κρατών μελών, αλλά για τη συνολικά, συνολική ευημερία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση, θα έλεγα. Ευχαριστώ. Mr. Κύριος Κρέστερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ για τα ενδιαφέροντα τα οποία μας εκθέσατε. Σε τρία σημεία να αναφέρω κάτι. Για το πρώτο, υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ τεχνικών και κοινωνικών καινοτομιών που θα μπορούν να την χάνουν κάλυψης από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Κανονικά για τεχνολογικές ή τεχνικές καινοτομίες γίνεται λόγος. Αλλά τι γίνεται με τις κοινωνικές καινοτομίες και αυτές μπορούν να καλυφθούν από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και ποιο είναι το ποσοστό μεταξύ τεχνικών και κοινωνικών καινοτομιών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Δεύτερο, για την υλοποίηση. Και όσον αφορά και την παραβίαση ή παράβαση των θεμάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που έχουν κατατεθεί σε εσά. Αν κάποιο έχει ένα δίπλωμα το οποίο έχει κατατεθεί σε εσά και κάποιο άλλο το μιμείται ή το αντιγράφει, ε, τότε πρόκειται για παραβίαση, έτσι δεν είναι, και ποια συνέχεια δίνεται. Και το τρίτο, κατάλαβα σωστά ότι σε σχέση με το TTIP, την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και Επενδύσεων, έχετε κάποιε επιφυλάξει όσον αφορά την διασφάλιση του δικαίου ε, το, της νομολογίας ε, των διπλωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όσον αφορά την οικονομική πτυχή. Ε, Κύριος Χρυσόγονος, παρακαλώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην Επιτροπή μας. Το άρθρο 30 των κανονισμών των διατάξεων για τις υπηρεσίες μονίμων υπαλλήλων του γραφείου σας προβλέπει ότι ο πρόεδρος μπορεί να καθορίσει όρους και διατάξεις για την άσκηση των δικαιωμάτων απεργίας ε, για τους υπαλλήλους σας. Και αυτοί οι όροι και διατάξεις ε, μεταξύ άλλων προβλέπουν και μια μέγιστη διάρκεια για τις απεργιών και τις ε, διαδικασίες ρύθμισης. Αυτά μου φαίνονται ότι περιορίζουν ε, δυσανάλογα τα δικαιώματα απεργίας ε, των υπαλλήλων σας. Εσείς ή το Διοικητικό Συμβούλιο συμβουλευθήκατε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας προτού να εγκρίνετε αυτές τις διατάξεις. Αναδείτε αν με, τις, ε, με τα άρθρα 87 και 98 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας είναι συμβατές οι δικές σας διατάξεις. Και πώς θεωρείτε το, την απόφαση του εφετείου στη Χάγη όπου αναφέρθηκε ότι παραβιάσεις του Διεθνούς εργασιακού, εργατικού δικαίου δεν μπορούν να δικαιολογούνται μονομερώς. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Καβαντά, παρακαλώ. C'est une erreur, Δεν ήθελα το λόγο. Λάθος. Νομίζω ότι έχω καλυφθεί. Ευχαριστώ. Ε, Mr. Anderson. Ο κύριος Άντερσον. Ja, ε, Eh, Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τον προσκεκλημένο μας για την εξαιρετική του παρουσίαση όπως την θεωρώ. Θα ήθελα μια ερώτηση να διατυπώσω για τις συμβουλές που θα μπορούσατε να μας δώσετε εσείς σε εμά τους πολιτικούς, τους ευρωβουλευτές. Τι μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε να αποφύγουμε μια ξεχωριστή ανάπτυξη του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών. Να μην μπορούν δηλαδή οι μεγάλες ε, επιχειρήσεις που έχουν μεγάλα τμήματα νομομαθών ε, να έχουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας αλλά έτσι να μπορούν να καταβυθίσουν τα συμφέροντα των μικρότερων. Τι θα μας ε, συμβουλεύατε σε σχέση με την κατάσταση όπου βλέπουμε στις ΙΠΑ ε, να υπάρχει, όπου γίνεται κατάχρηση των συστημάτων ευρεσιτεχνίας. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια εξέλιξη και μια τέτοια κατάσταση. Τι θα μας συμβουλεύατε. Ευχαριστώ. Αυτοί ήταν οι αγορητές που ζήτησαν να παρέμβουν. Κύριε Πρόεδρε, έχετε και πάλι τώρα τον λόγο, παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στα γαλλικά. Πάλωστε είναι μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Απευθυνόμενος καταρχάς τον κύριο Φως, να πω ότι σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας, για την λύση αυτή την οποία προβλέπουμε, τις τέσσερις αυτές πρώτες λύσεις όσον αφορά το ζήτημα των τελών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθεί μία ισορροπία ανάμεσα σε τρεις συγκεκριμένες δυσκολίες που υπάρχουν. Πρώτον, το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνία θα πρέπει να είναι ελκυστικό για τις επιχειρήσεις, business attractive όπως λέμε στα καλά γαλλικά. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία, διότι το δίπλωμα αυτό, το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία, απευθύνεται τελικά σε 27 χώρες του οι υπόλοιπες 13 που δεν εντάσσονται στο σύστημα αυτό, θα πρέπει να συνειδητοποιούν βέβαια ότι το παγκόσμιο σύστημα χρηματοδοτεί το ενιαίο δίπλωμα βρεστεχνία. Χρειαζόμαστε λοιπόν να κρατήσουμε μια κάποια δημοσιονομική ισορροπία και ουδετερότητα. Και τέλος, θα πρέπει να δημιουργούμε κάποιους πόρους, κάποια έσοδα για τα κράτη-μέλη προκειμένου να μπορούν και αυτά να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πολιτική τους, ιδίως όσον αφορά την ευαισθητοποίηση εκείνη για την καινοτομία και για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πάντως, νομίζω ότι ο πρώτος στόχος που ανέφερα είναι ο πιο σημαντικό από τους τρεις και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήρθαμε σε ευρία διαβούλευση με όλους ενδιαφερόμενους φορείς, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πελατών, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή. Πελάτες οι οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρώπης και θεωρώ ότι η πρόταση αυτή που έκανα θα πρέπει τελικά να προσελκύσει και μία ευρεία υποστήριξη, διότι αποτελεί την κατάλληλη ισορροπία δίνοντας προτεραιότητα σε οικονομικές επιπτώσεις. Να απευθυνθώ τώρα στην ερώτηση του κυρίου Κλάστερ. Μόνο οι τεχνικές καινοτομίε είναι αυτές οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Πολύ συχνά λέμε ότι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποτελεί μια τεχνική λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα. Συνεπώς, οτιδήποτε δεν διαθέτει αυτή τη τεχνική διάσταση βρίσκεται εκτός πεδίου εφαρμογής του, διπλωμα, του διπλώματος Οι κοινωνικές, για παράδειγμα, καινοτομίε, οι καινοτομίε σε άλλου τομεί, οι ιδέε οι ίδιε δεν μπορούν να καλυφθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Ο δικός μας ο τομέας λοιπόν είναι πολύ σαφώς οριοθετημένος και απευθύνεται όπως σας είπα στις βιομηχανικές εκείνες διαδικασίες οι οποίες όλο και περισσότερο καλύπτουν βέβαια και την ψηφιακή οικονομία, αλλά και πολλές ψηφιακές υπηρεσίες. Πάντως το γενικότερο πλαίσιο παραμένει ένα πλαίσιο που αφορά τις τεχνικές καινοτομίες. Επίσης και έχετε απόλυτο δίκιο που το αναφέρατε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κατοχυρώνουμε διπλώματα βραστιτεχνίας, να κατοχυρώνουμε δικαιώματα, αν αυτά στην πράξη δεν τηρούνται. Δυστυχώ όμω το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά την επιβολή των διπλωμάτων, διπλωμάτων και την επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων. Είμαστε ένα οργανισμό με σαφεί αρμοδιότητε, αρμοδιότητε που μα έχουν παραχωρήσει τα κράτη-μέλη και περιορίζονται στην ε, κατοχήρωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στη δημιουργία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ε, προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, οτιδήποτε έχει να κάνει με την καταπολέμηση της απάτης, της απομίμησης κτλ, της παραποίησης, όλα αυτά αποτελούν αρμοδιότητες που είναι κυρίως εθνικές και σε ορισμένες περιπτώσεις ευρωπαϊκές. Όσον αφορά τώρα το TTIP, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έλλειψη ισορροπίας στις συζητήσεις. Δηλαδή από τη μία πλευρά έχουμε την Αμερικανική αντιπροσωπεία η οποία έχει πολύ συγκεκριμένε ιδέες για πολύ συγκεκριμένα σημεία όσον αφορά τη διαδικασία διπλώματος ευρεσιτεχνίας και από την άλλη έχουμε την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει την ίδια τεχνική και νομική αρμοδιότητα με τις ΗΠΑ σε αυτό το τομέα. Πρώτον αυτό. Επομένως, ας είμαστε πολύ προσεκτικοί Πολλές φορές στα πλαίσια των συζητήσεων ε, ορισμένα ζητήματα τα θεωρούμε ίσονος σημασίας, όπως για παράδειγμα η χρονική περίοδος, η περίοδος χάριτος η λεγόμενη. Ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός όσον αφορά τα συστήματα διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Λέμε ότι ο εφευρέτης είναι ο πρώτος ο οποίος υποβάλλει ένα αίτημα κατοχήρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, δεν ισχύει μόνο αυτό το απλό κριτήριο, θέλουν να δουν πραγματικά ποιος είναι ο πραγματικός εφευρέτης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχουν πάρα πολλές προσφυγές που μπορούν να προκύψουν και καλούμεθα εμείς να επιλύσουμε πάρα πολλές διαφορές για να καταφέρουμε να καταλήξουμε στον πραγματικό εφευρέτη κάθε φορά. Ορισμένα πράγματα φαίνονται εκ πρώτης όψεως απλά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ευρωπαϊκής και αμερικανικής νομοθεσίας και ενδεχομένως δεν είναι στα πλαίσια του τύπου που θα πρέπει να επιληθούν οι διαφορές αυτές. Κύριε Χρυσόγονε, εσείς αναφερθήκατε στο δικαίωμα απεργίας και υποβάλλετε ένα σχετικό ερώτημα. Πρέπει να σας πω ότι όντως στα πλαίσια των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που αφήρμοσα για πρώτη φορά αναγνώρισε το δικαίωμα απεργίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Δεν αναγνωριζόταν στο ΕΠΙΟ το δικαίωμα αυτό στο παρελθόν και είναι σαφώς οριοθετημένο το δικαίωμα αυτό, δηλαδή διέπεται από συγκεκριμένου κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους η απεργία θα πρέπει να αποτελεί ίστατο μέσο όσον αφορά τις κοινωνικές αυτές εργασιακές σχέσεις. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς και καταχρηστικά το δικαίωμα αυτό αλλά μόνο σε περίπτωση κατάρρευσης και αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να πω επίσης ότι στα κράτη-μέλη τα οποία παρτίζουν το EPO υπάρχουν ορισμένες χώρες που δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα απεργίας των υπαλλήλων. Εγώ όμως, ανταυτού, αναγνώρισα το δικαίωμα απεργίας για όλους προφανώς εργαζομένους, για όλους υπαλλήλους του EPO, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Τώρα, όσον αφορά το Διοικητικό Δικαστήριο του ILO, Προφανώς εμείς έχουμε εμπνευστεί από τους κανόνες και τις βασικές αρχές του οργανισμού αυτού, αρχές που δημοσιεύει αυτός ο οργανισμός και πρέπει να σας πω ότι, το, ότι γίνονται πολλές προσφυγές κατά του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρωστεχνίας και θα έλεγα ότι ένα 90-95% των προσφυγών αυτών εκδικάζονται από το δικαστήριο αυτό. Και πέρυσι, δυστυχώς, είχαμε 22 μέρες απεργίας στις οποίες συμμετείχαν μόνο 12% των υπαλλήλων. Όσον αφορά τώρα την απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης, είμαστε ενώπιον μιας κατάστασης όπου μια εθνική δικαιοδοσία δεν θεωρείται αρμόδια προκειμένου να εκδικάσει τον τρόπο διοργάνωσης ενός διεθνούς οργάνου. Αν μια εθνική δικαιοδοσία, για παράδειγμα, επενέβαινε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ αυστηρό όσον αφορά την, τις αρχές τις οποίες θα πρέπει να διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι όλα τα δικαιώματα της ασυλίας τα οποία προβλέπονται για τον EPO έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν την αυτονομία και την εξαρτησία του EPO. Έχουμε λοιπόν μία απόφαση η οποία έχει ένα μοναδικό ξεχωριστό χαρακτήρα. Ξέρετε ότι γίνανε πάρα πολλές προσφυγές στο παρελθόν που μας είχαν δικαιώσει. Θεωρώ ότι έχει γίνει ένα λάθος λοιπόν από το δικαστήριο αυτό και βλέπουμε ότι και η ίδια η κυβέρνηση των κάτω χωρών μας υπεράσπισε στην έφεση που κάναμε κατά της απόφασης αυτής ε, του δικαστηρίου. Πρέπει να σας πω επίσης ότι το κοινωνικό πακέτο, η κοινωνική δέσμη την οποία παρέχουμε στο ΕΠΟ είναι ιδιαίτερα γενναιόδορη. Σας καλώ πραγματικά να συμβουλευτείτε την κοινωνική έκθεση την οποία δημοσιοποιούμε κάθε χρόνο και είμαι ο πρώτος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ο οποίος σε τήσια βάση κοινοποιεί τέτοια διαφανή και λεπτομερή έκθεση όσον αφορά τη μισθοδοσία, όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, όσον αφορά το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, όσον αφορά τα δικαιώματα φροντίδας των παιδιών, όσον αφορά το δικαίωμα στις διακοπές που έχουν οι υπάλληλοι μας. Θα δείτε λοιπόν, αν διαβάζετε την έκθεση αυτή, ότι το κοινωνικό μας σύστημα είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο και είμαι υπερήφανος που φτάσαμε στο επίπεδο αυτό, αλλά είναι σημαντικό να καταφέρνουμε και μακροπρόθεσμα να χρηματοδοτούμε αυτό το γενναιόδωρο σύστημα, γιατί αν δεν καταφέρουμε να το κάνουμε εμείς, είναι τα κράτη-μέλη που θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν την κοινωνική μας αυτή πολιτική. Η πολιτική λοιπόν που εγώ εφαρμόζω στον οργανισμό αυτό έχει ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητά μας, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά μας, προκειμένου μας σε θέση και στο μέλλον να παρέχουμε τις ίδιες ποιοτικέ υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο απλώς να αυξάναμε τα τέλη μας, να αυξάναμε τις τιμές μας. Δεν θα κάναμε τίποτα ουσιαστικό και απλώς θα αυξάναμε τις τιμές μας. Δεν νομίζω όμω ότι κάτι τέτοιο περιμένει από εμάς η ευρωπαϊκή οικονομία. Τέλος, κύριε Άντερσον, Πιστεύω ότι αυτό που προσάπτουμε στο γενικότερο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν έχει τόσο σχέση με τους κανόνες και τις αρχές, αλλά κυρίως με την δυσλειτουργικότητά του. Και ειλικρινά σας το λέω, το λέω ανοιχτά, ότι αυτό προκύπτει πολύ πιο συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι τόσο στην Ευρώπη. Πολύ περισσότερες είναι οι ενστάσεις και τα παράπονα τα οποία εκφράζονται στις Ηνωμένες και όχι τόσο στην Ευρώπη. Συνεπώς, θεωρώ ότι στην Ευρώπη έχουμε κάποιους καλούς κανόνες. Πρώτον, και βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχει και μια διαφορά νοοτροπίας. Το Αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία κατοχυρώνει με διπλώματα ευρεσιτεχνία πολύ πιο εύκολα και γρήγορα από ότι το EPO και υπάρχουν τελικά πάρα πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνία τα οποία αναγνωρίζονται τελικά στι ΗΠΑ χωρί να χαίρουν αναγνώριση όμω στην Ευρώπη και οι Αμερικάνοι ακολουθώντας το γενικότερο σύστημα το οποίο έχουν θεωρούν ότι θα πρέπει τα δικαστήρια να αποφανθούν στη τελική ανάλυση. Εμείς στην Ευρώπη θεωρούμε ότι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι πιο αυστηρό, πιο επιλεκτικό προκειμένου να έχουμε λιγότερο, λιγότερες δικαστικές διαμάχες. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε εθνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή, σε εθνικές δικαιοδοσίες στην Ευρώπη έχουμε λιγότερες νομικές διαφορές και λιγότερε δίκε εκδικάζονται όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Θεωρώ λοιπόν το δικό μα το σύστημα με του κανόνε που έχει είναι πολύ πιο ισορροπημένο. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε βήμα-βήμα τελικά μεταρρυθμίζουν το δικό του σύστημα και προσεγγίζουν περισσότερο το δικό μα το ευρωπαϊκό σύστημα. Και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό και θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη παγκόσμια ισορροπία όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Και άλλωστε και η ίδια Ευρώπη θα πρέπει να είναι περήφανη που χρησιμοποιεί αυτό το λεγόμενο soft power προκειμένου να καταφέρει να προσελκύσει και άλλες χώρες και συγκεκριμένα και τις ΗΠΑ προς το δικό της το σύστημα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ελπίζω να απάντησα σε ερωτήσεις. Uh, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που απαντήσατε στις ερωτήσεις. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητά το λόγο. Δεν θέλει κανείς άλλος να σας θέσει ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για το χρόνο που αφιερώσατε και για την επίσκεψη στην Επιτροπή μας. Δεν καλωσόρισα τους συναδέλφους σας που βλέπω εδώ στην αίθουσα. Να τους αποχαιρετήσω τουλάχιστον και να αποχαιρετήσω και εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας στη διάρκεια της ε, συνεχούς μας ε, συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. everybody's in place, so we can continue, I guess. So, we may... Λοιπόν, να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι. Επόμενο σημείο, το σημείο παριθμών 5, η ακρόαση για το ζήτημα των ευρωπαϊκών ελάχιστων προτύπων για την πολιτική δικονομία. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, ε, Μπούρκαντ Χες, τον εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Max Planck ε, στο Λουξεμβούργο και την κυρία Εύα Στρόσκρουμπ, ε, με συγχωρείτε για τον τρόπο που προφέρω το επιθετό σας από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλλας, καθώς επίσης και την ε, γνωστή προσκεκλημένη μας, την Ταϊάννα Γουόλης, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Νομικής και τον Μάικλ Σότερ, επικεφαλής του Τμήματος ε, Πολιτικής Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας καλωσορίζω όλους και θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Χέση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, την παρουσίασή μου την έχω προετοιμάσει στα αγγλικά θα σας την παρουσιάσω όμως στα γερμανικά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Το θέμα μου είναι η σύγκληση των δικονομικών ε, δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Και θα ξεκινήσω μιλώντας για την κατάσταση που έχουμε σήμερα μπροστά μας στην Ευρώπη. Βλέπετε σε αυτό το γράφημα το Judicial Scoreboard, τον πίνακα επιδόσεων και τις διαφορετικές επιδόσεις των συστημάτων αστικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε πραγματικά καθοδόν προς την σύγκληση των δικονομικών δικαιωμάτων. Όμως οι διαφορετικές, ας το πω έτσι, ικανότητες και δυνατότητες ε, των αστικών συστημάτων στην Ευρώπη δεν βασίζονται μόνο φυσικά σε διαφορετικά δικονομικά δικαιώματα και δυνατότητες αλλά σε διαφορετικές δομές ε, των ε, συστημάτων ένα θέμα το οποίο όλο και περισσότερο αποκτά τη σπουδαιότητά του. Ο ρόλος των δικαστών και των ε, ως εμπλεκόμενων μερών είναι διαφορετικός ο ρόλος αυτός και τα διαφορετικά διαδικαστικά δικαιώματα. Και ένα σημαντικό θέμα και γι' αυτό σε, αυτό το, σε αυτή τη διαφάνεια που σας δείχνω βασίζεται και στη διαφορετική χρηματοδότηση των δικαστικών συστημάτων, ε, δικονομικών συστημάτων στα κράτη-μέλη περίπου μπορούμε να διακρίνουμε ότι ε, με, συγκρίνοντας με την πρώτη διαφάνεια πόσο διαφορετικά χρηματοδοτούνται τα δικαστικά συστήματα. Όσο σκουρότερο είναι το χρώμα, όσο πιο σκούρο πράσινο είναι το χρώμα, τόσο καλύτερα είναι αυτά τα συστήματα όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους. Επικεφαλής είναι το Λουξεμβούργο αυτό δημιουργεί κάποια μηχανία για μένα. Έχουμε υψηλότερο ποσοστό ε, πολίτη για την εισφορά. Κατεβαίνουμε στα 32 ε, βλέποντας ε, την ε, ε, γειτονική χώρα. Και έχουμε εδώ τις διαφορετικές επιδόσεις των δικαστικών συστημάτων. Το Λουξεμβούργο <clears throat> βρίσκεται πολύ μπροστά στις επιδόσεις. Πρώτο κράτος. Η Γαλλία πληρώνει 61 ευρώ βρίσκεται όμως ετήσια 61 ευρώ βρίσκεται όμως περίπου στην ίδια γραμμή όπως, όσον αφορά την αποδοτικότητα όπως η Ισπανία. Στην Ισπανία αποφασίζουν 10 δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο για όλα τα, όλες τις αστικές υποθέσεις ε, της χώρας. Στην Γερμανία είναι 92 δικαστές ε, που αποφασίζουν σχετικά. Στην Ισπανία έχουμε περίπου 42 εκατομμύρια πολίτες, στη Γερμανία 80 εκατομμύρια πολίτες. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν για ποιο πράγμα κάνουμε λόγο εδώ και πώς όλα αυτά ε, μπορούν να αντιμετωπιστούν σε ένα ιστό. Πρόκειται για τον συντονισμό αλλά και τον ανταγωνισμό μεταξύ τους των διαφορετικών δικονομικών συστημάτων από πλευρά δικαιοσύνη. Θα ήθελα εδώ δύο προοπτικέ να καταδείξω. Αφενό την προοπτική του ενωσιακού δικαίου, αφετέρου την προοπτική του δικαίου των κρατών μελών. Υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, το θέμα είναι η δικαιοσύνη να μπορεί να είναι αποδοτική για την ενιαία εσωτερική αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Διασυνοριακά να μπορούν να συντονίζονται και να επιλύονται διαφορές. Και ο συντονισμός όπως γνωρίζετε λειτουργεί μέσω διαφορετικών μέσων που ξεκινούμε με τον κανονισμό 1 διαδικαστικά είναι ένας απλός κανονισμός σχετικά που ε, στοχεύει στο να επιτευχθεί ουσιώδης συντονισμός. Έχουμε όμως και πολύ διαφορετικά μέσα. Ένα από τα πιο πρόσφατα είναι ο κανονισμός για την ε, ε, ευρωπαϊκή ε, λειτουργία των, λογαριασμών. Προβλέπεται εξειδικευμένη ρύθμιση που θέτει και ελάχιστες προδιαγραφές ελάχιστες προδιαγραφές ως στάνταρς Βρισκόμαστε ακριβώς στο θέμα. Κατά πόσο χρειάζονται στην Ευρώπη τέτοιες ελάχιστες προδιαγραφές ε, διαδικαστικά. Από πλευράς Λένατς ε, στην Oxford ε, παρουσιάστηκε μια σημαντική παρέμβαση όσον αφορά την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Είπε ο Λένατς ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη στα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών μπορεί μόνο τότε να λειτουργήσει όταν, και το αναφέρω αγγλικά, μπορεί να διευρύνει την νομοθεσία. Δηλαδή όταν η νομοθεσία το νομοθετικό πλαίσιο μέσω διαδικασιών, διαδικασιών εφαρμοστικών μπορεί να λειτουργεί. Και έχει δίκιο σε αυτή την άποψή του. Χωρίς τέτοιου είδους ε, διατάξεις ε, που θα μπορούν να διασφαλίζουν την ε, αποτελεσματική διανομή των εγγράφων και την αμεροληψία μπορούμε όταν λειτουργούμε έτσι να έχουμε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως προς αυτό. Έχουμε την προοπτική λοιπόν, μια στιγμή κάτι δεν πήγε καλά, των κρατών μελών. Ψάχνει τη διαφάνεια ο μιλητής. Μια ακόμα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφάνεια, η σωστή διαφάνεια. Για τα κράτη-μέλη τώρα. Το πρώτο βήμα ποιο είναι. Και εδώ υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα <clears throat> να μπορεί να εφαρμόζεται σωστά το δικονομικό πλαίσιο, το διαδικαστικό πλαίσιο. Κανονισμοί μέσω συνοδευτικών μέτρων να μπορούν να προωθούνται στα εθνικά συστήματα και να μεταφέρονται και να εκτελούνται σε αυτά. Για τον κανονισμό Βρυξελών 1α που εφέτος άρχισε να λειτουργεί αυτό είναι κέρια σημασία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει τα κράτη-μέλη πραγματικά να αναλαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα και διαβήματα για να προχωρήσουμε. Τα κράτη-μέλη από πλευρά του έχουν σαφή ανταγωνισμό που ανέπτυξαν μεταξύ των εθνικών συστημάτων. Πρόκειται για έναν ανταγωνισμό λοιπόν εδώ μεταξύ εθνικών αγορών. Αγορών για νομικές υπηρεσίες. Όταν έχουμε το παράδειγμα financial litigation, μπορείτε να δείτε ότι οι οικονομικές τέτοιες διαφορές μεγάλου εύρους, μεγάλης εμβέλειας, μέσω συμφωνιών δικαστικών μπορούν να διευθετούνται litigation λοιπόν που μπορεί να λειτουργήσει στο Düsseldorf εν μέρη στην Ολλανδία ή και στην, ε, ε, στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ε, ενιαία εφαρμογή του κανονισμού Βρυξελών 1α, οι διαδικαστικές διαδικασίες διευκολύνουν τα πράγματα και ο ανταγωνισμός έτσι έχει αυξηθεί μεταξύ αυτών των εμπλεκομένων. Αυτό δεν είναι αρνητικό, μπορεί να οδηγήσει σε καινοτομίες και εξυγχρονισμό αλλά καμιά φορά παρακάμπτονται οι κανόνες και οι διατάξεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα είχαμε το νέο κανονισμό φερεγγιώτας ή πτώχευσης. Υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός στην Ευρώπη όσον αφορά την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και τις σχετικές διαδικασίες. Εδώ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό το αγγλικό πρότυπο προσέγγισης. Δυστυχώς ο κανονισμός ο κανονισμός ε, ε, πτώχευσης ε, καθορίζει σε ένα παράτημα τα σχετικά. Στο παράτημα τι βρίσκει κανείς. Βρίσκει τις εθνικές διατάξεις που εντάσσονται ή θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτόν τον κανονισμό προς εκτέλεση. Όταν τα κράτη-μέλη δεν αναφέρουν σχετικά μέσα, τότε δεν εντάσσονται, δεν υπάγονται σε αυτόν τον κανονισμό. Αυτό συμβαίνει σε αυτό το scheme arrangement. Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει ένα opt-out, μια εξαίρεση, αυτοεξαίρεση από αυτά τα ευρωπαϊκά νομικά μέσα. Πρέπει να μεριμνήσουμε, είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν στο πώς θα λειτουργήσουμε. Περνάω στο επόμενο βήμα, δηλαδή στο περαιτέρω πεδίο εφαρμογής ε, αυτών των διατάξεων. Αυτό αφορά την συγκυρία όπου επί της ουσίας το ευρωπαϊκό δίκαιο θα εφαρμόζεται. Ευρωπαϊκό καταναλωτικό δίκαιο έναντι εθνικών δικαίων που θα πρέπει να επικρατεί και να εφαρμόζεται. Και εδώ ισχύει η αρχή ότι κάθε δικαστήριο είναι ένα αποκεντρωμένο ενωσιακό δικαστήριο. Εφαρμόζουν το δικό τους διαδικαστικό δίκαιο τα δικαστήρια δικονομικά είναι, έχουν αυτή την αυτονομία στα κράτη-μέλη, όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ελέγχει πώς, πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται εθνικά όλα αυτά μέσα από την αμοιβαιότητα και αποτελεσματικότητα. Κυρίες και κύριοι, και τα δύο αυτά μέσα δεν είναι καθόλου ακριβή. Και πρέπει να πούμε ότι οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν μπορεί να προβλεφθούν ε, οι ε, περαιτέρω διατάξεις. Γι' αυτό υπάρχει ένα περαιτέρω πεδίο το οποίο πρέπει να αναμένουμε περισσότερα και είναι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο άρθρο 47 προβλέπει διαδικασίες εγγυήσεις που μπορούν να θεωρηθούν ως ελάχιστα εχέγγυα, ως ελάχιστες ε, εγγυήσεις. Όταν πάντα επί της ουσίας εφαρμόζεται ενωσιακό δίκαιο, τότε η ελάχιστη εγγύηση από πλευρά τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ισχύει. Σας δίνω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Το εφετείο στην ε, ε, Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε για μια προσφυγή. Ε, χρήστες υπολογιστών Apple χρησιμοποιούσαν ένα ψαχτήρι, browser, που είχε όμως ε, ε, χρησιμοποιούσε διαφημίσεις στοχευμένα ώστε να περάσουν οι διαφημίσεις στους χρήστες αυτού του ψαχτηριού. Αντέδρασαν οι χρήστες κατά αυτών των ε, διαφημίσεων. Το θέμα που τέθηκε στο εφετείο, το βρετανικό εφετείο ήταν θα υπάρχουν αποζημιώσεις για μη υλικές ζημιές μπορούν να απαιτηθούν. Σύμφωνα με την, ε, το εφαρμοστικό δίκαιο στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με την οδηγία προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ήταν δυνατό να γίνει αυτό. Όμως το δικαστήριο αναφέρθηκε στο άρθρο 47 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και είπε πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας και γι' αυτό ήταν παραδεκτή η προσφυγή. Αυτό δείχνει ποια αποτελεσματικότητα έχει η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και πώς μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά αποτελεσματικά. Προ αυτού του κοινικού τίθεται το ερώτημα τι γίνεται σε σχέση με τη σύγκληση όσον αφορά τα νομικά πλαίσια. Και εδώ υπάρχουν φυσικά διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές δυνατότητες. Αυτές οι διαφορετικές δυνατότητες και προσεγγίσεις έχουν τύχει χρήσης μέχρι σήμερα. Η πρώτη προσέγγιση σε διαφορετικούς τομείς εξειδικευμένες νομικές πράξεις μπορούν να εκδίδονται. Υπήρξαν τέτοιες πράξεις. Για παράδειγμα, <clears throat> είχαμε την ε, ευρωπαϊκή ε, ρύθμιση όσον αφορά λογαριασμούς. Και βλέπουμε εδώ ότι αντανακλώνται ελάχιστες προδιαγραφές πάλι. Προδιαγραφές που προβλέπουν ένα ελάχιστο διαδικαστικό επίπεδο προστασίας. Έχουμε παράλληλα ξεχωριστές διαδικασίες. Η πιο περιβόητη διάταξη είναι η διάταξη ε, για, για τις προσφυγές περίπου 500, 500 έως 600 τέτοιες προσφυγές έχουμε στη Γερμανία με βάση αυτό το δίκαιο. Έχουμε 1,2 εκατομμύρια έναντι των ε, ε, πρωτοδικείων για παράδειγμα και βλέπουμε ότι υπάρχει μια παρέκκληση όσον αφορά αυτές τις ε, ρυθμίσεις. Δεύτερον, ένα ενιαίο πλαίσιο για την διευθέτηση διαδικασιών Έχουμε το Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Γραφείο τεχνιών, Το εξετάσατε αυτό το θέμα. Και υπάρχει και η δυνατότητα να υπάρχουν μη δεσμευτικέ συστάσει και μέσω αυτών να προετοιμάζονται περαιτέρω νομικέ πράξει. Παράδειγμα, η σύσταση για την συλλογική προστασία που σίγουρα σε ένα δεύτερο βήμα θα οδηγήσει σε περαιτέρω λήψη νομικών μέτρων και εφαρμογή τους. Και ένα άλλο παράδειγμα είναι η πρόταση που αφορά το Ευρωπαϊκό Νομικό Ίδρυμα ώστε να υπάρξει ένα πρότυπο νομικό, υπόδειγμα νομικό για, την, για τα αστικά δικαστήρια μέσα στο πλαίσιο του αστικού δικαίου. Αυτά είναι τέτοιου είδους μέτρα ως παραδείγματα που είναι ενδιαφέροντα διότι αντανακλούν την ε, αποδεκτικότητα, την αποδοχή τους. Γιατί να ρυθμίζονται τα δικονομικά, τι εξυπηρετείται η εξαπλούστευση και μόνη της, από μόνη της δεν μπορεί να επαρκεί και να δικαιολογεί τις διαδικασίες. Ένα ουσιώδες στοιχείο και αυτή είναι η ευκαιρία της Ευρώπης είναι οι εθνικές διαδικασίες να εξυγχρονιστούν, να μεταρρυθμιστούν όπου είναι αναγκαίο να γίνει αυτό. Παράδειγμα, e-justice, ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Παράδειγμα, βελτίωση όσον αφορά τις ε, ε, διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης ε, διαδικασιών IP. Εξάλλου, ισότητα ευκαιριών που πρέπει να διασφαλίζεται για τους οικονομικά εμπλεκόμενους και τις επιχειρήσεις. Σημαντική πτυχή αυτή θα πρέπει ε, να αποφύγουμε μακροπρόθεσμα στρεβλώσεις ή υπονόμευση. Στόχος πρέπει να είναι η πρόσβαση των πολιτών να διασφαλίζεται σε αυτά τα ανεμικά πλαίσια. Και πρέπει να προσέξει κανείς και το λέω αυτό ανοιχτά και αθυρόστομα ώστε μέσω εναλλακτικών συστημάτων να μην ε, παρακολύεται ο πολίτης αντί να διευκολύνεται στο να διασφαλίσει την προσπελασιμότητά του σε αυτά τα συστήματα. Και εδώ πρόκειται επίσης για την ενδυνάμωση της οικονομίας. Όχι για τα θέματα πτώχευσης αλλά και για τα θέματα της της διαδικασίας της Τρόικας, της Τριμερούς, στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία είχαμε ευρύτερες και σημαντικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα δικαστικά συστήματα και σε πλαίσιο με την οικονομική κρίση. Τώρα, τι θα έπρεπε να είναι η σωστή, ποια θα έπρεπε να είναι η σωστή στρατηγική, ώστε διαδικαστικά να μπορούν να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Αφενός πιστεύω ότι μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνάφεια είναι σίγουρα αναγκαία, διότι στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές φορές ε, τομεακά εξειδικευμένα πρέπει να αντιμετωπίζονται συγκεκριμένα προβλήματα. Και ίσως η ιδέα ενός ολοκληρωμένου ε, συνολικού συστήματος ίσως μπορεί να απολεστεί. Πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε κατά πόσον μπορούμε να πάμε πιο πέρα ή όχι. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Οι μακρότατες συζητήσεις για ένα ενιαίο συμβατικό δίκαιο όσον αφορά το αστικό πλαίσιο, τον, ε, τον αστικό τομέα δείχνει το τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνετοί και προσεκτικοί, αλλά μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνοχή είναι σίγουρα σημαντικό στοιχείο μεγαλύτερη καινοτομία όσον αφορά αυτές τις διαδικασίες είναι αναγκαία. Και θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει προχωρήσει σε αυτόν τον τομέα για τη διαμεσολάβηση για παράδειγμα. Όσον αφορά συλλογικές ε, υποθέσεις πρέπει τουλάχιστον διασυνοριακά τα μέσα αυτά να μπορέσουν να καταλήξουν σε ένα μέσο το οποίο θα είναι αποτελεσματικό. Και e-justice είναι σίγουρα η ηλεκτρονική δικαιοσύνη το, μέτρο, το μέσο εκείνο για να μ, καινοτομήσουμε και να μεταρρυθμίσουμε τα ανεδαφικά ή ε, μη αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα. Καθώς επίσης και μέσα όπως ε, συστάσεις ε, που πρέπει να μπορέσουν να δημιουργήσουν δυνατότητες που θα αντικατασταθούν στη συνέχεια μέσω νομικών πράξεων. Όσον αφορά για παράδειγμα τις εξοδικαστικές ε, ε επιλύσεις ε, ε, αντιπαραθέσεων. Οι συστάσεις όμως αυτές θα πρέπει να γίνονται, να είναι πιο συστηματικές, να είναι καλύτερες, καλύτερης ποιότητας. Δεν μπορεί απλά και μόνο να είναι μια εργαλειοθήκη, ένα toolbox που θα διατίθεται στα κράτη-μέλη. Πρέπει να μπορούμε να δημιουργούμε τη βάση για τις νομικές πράξεις που συστηματικά θα προετοιμάζονται. Ελάχιστες προδιαγραφές. Σίγουρα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να οδηγηθούμε σε μια ουσιώδη μεταρρύθμιση των συστημάτων αυτών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ζητώ συγγνώμη που πρέπει να αποχωρήσω νωρίτερα, διότι έχω υποχρεώσεις ανηλυμένες και πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much, Professor Hess. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά Χες. Να δώσω τώρα το λόγο στην Εύα Στόρσκουπ από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλλας. Um, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ για να μπορέσουμε να σας απευθύνω το λόγο για το θέμα αυτό. Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ με τον ε, καθηγητή Χέσ και την Ταϊάννα Γουόλης. Το θέμα το οποίο μου δόθηκε είναι η δημιουργία κοινών προδιαγραφές ε, κοινής δικονομίας ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αποφάσισα να το χωρίσω σε τρεις ενότητες. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το τέλος. Καταρχάς θα αναφερθώ στη ε, πολιτική δικονομία στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τι είναι. Μετά θα ξεκινήσω τις κοινέ προδιαγραφές, ε, τι είναι οι κοινέ προδιαγραφές. Και τέλος, όταν θα συζητήσουμε τη δημιουργία των κοινών προδιαγραφών, θα ε, συζητήσουμε τι ακριβώς είναι αυτή η δημιουργία. Πρέπει να σας πω ότι στις διαφάνειές μου χρησιμοποιώ τον όρο «εμείς». θα μπορούσε βέβαια κάλλιστα αυτό το «εμείς» να είναι ένα ουδέτερο ε, πρόσωπο, αλλά χρησιμοποιώ αυτό το εμείς, διότι αναφέρομαι σε μας, εμάς εδώ το, σήμερα, αλλά και τον ευρύτερο κλάδο των νομικών, των νομοθετών, ε, των ανθρώπων που ασκούν ε, τη νομική, που συμμετέχουν στην πρόοδο και στην εξέλιξη της πολιτικής οικονομίας στην Ευρώπη. Τι εννοούμε με τον όρο πολιτική δικονομία. Ο καθηγητής Χέι αναφέρθηκε ήδη σε πολλά από τα θέματα τα οποία θα αναφέρω εν συντομία εγώ εδώ σήμερα. Στην Ευρώπη υπάρχει ένα πολύ ε, ποερίπλοκο, πολυεπίπεδο σύστημα και έχουμε μία εικόνα τι, τι θα μπορούσε να είναι πολιτική δικονομία σήμερα. Φανταστείτε ότι έχουμε ε, συνεργασία σε αστικά ε, θέματα ε, θα θυμα... γνώριζε το άρθρο 91 που αποτελεί τη βάση για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών και όπως ανέφερε και ο καθηγητής ε, Χες, σήμερα πλέον υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε διαδικασίες οι οποίες εκπονούνται βάση της πολιτικής οικονομίας. Η πιο πρόσφατη είναι το Ευρωπαϊκό Έντελμα Διατήρησης Λογαριασμών. Ε, αυτό Βέβαια, θα πρέπει, να το έχουμε, που ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι αφορά καθαρά διασυνοριακά ζητήματα και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία έχουν συγκεκριμένη θέση από τα, ε, επί των θεμάτων αυτών και δεν θα πρέπει να το λησμονούμε όταν αναφερόμαστε σε κοινέ προδιαγραφές. Επίσης, ε, έχουμε το συγκεκριμένο κλάδο που ανέφερε και ο κύριος Χέ, αυτό που αποκαλώ εγώ συγκεκριμένη νομοθεσία ένα κλάδο και υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρουσε νέε εξελίξει στα θέματα καταναλωτικού δικαίου, δικαίου ε, πνευματικών δικαιωμάτων και δικαίου ανταγωνισμού, αλλά αυτέ οι εξελίξει είναι τόσο πρόσφατε, που κανένα από τα στοιχεία που θα αναφέρω στη διαφάνεια δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ. Είτε θα τεθούν σε ισχύ του χρόνου, είτε ε, το 2017. Επομένω, δεν θα γνωρίζουμε επακριβώ τι θα σημαίνει αυτό για την πολιτική δικονομία στην Ευρώπη ακόμα. Επίσης υπάρχει αυτό το οποίο πολύ συχνά αποκαλείται ε, το δόγμα ε, της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με την ισοδυναμία και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και κυρίως το σκεπτικό ότι ε, υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματική αποζημίωση όταν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δικαίωμα που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και μετά έχουμε το συνταγματικό επίπεδο, το άρθρο 47 της ε, συνθήκη ω τέταρτο σκέλο. και το πέμπτο σκέλο είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να πολύ συχνά λησμονείται. Είναι μια πληθώρα μέτρων που προσπαθούν να έχουν ε, γενικότερες συνέπειες ε, στο σύστημα αστικής δικαιοσύνης. Ένα πρόσφατα ε, νέο στοιχείο είναι οι πίνακες επιδόσεων της δικαιοσύνης, καθώς επίσης και μία απόπειρα που γίνεται για τη δημιουργία ε, δικτύων μεταξύ δικαστών ή άλλων ατόμων που ασκούν ε, ε, νομικά επαγγέλματα, κάτι το οποίο λειτουργεί σε κάποιο βαθμό. Έχουμε λοιπόν πέντε βασικά παρακλάδια και όταν αναφερόμαστε σε κοινέ προδιαγραφές στην ευρωπαϊκή πολιτική δικονομία, θα πρέπει να λάβουμε και αυτά τα πέντε παρακλάδια υπόψη και να δούμε τι σχέση έχουν μεταξύ τους. Ε, ελοχεύει βέβαια ο κίνδυνο να θεωρηθεί μια εξέλιξη η οποία ε, είναι εμβαλωματική, κάτι το οποίο συμβαίνει ε, σκόρπια. Ε, κάτι όμως ε, το οποίο θα μπορούσε κάποιος προβληματικό, θα μπορούσε ίσως και κάποιος να θεωρήσει ότι αναπαράφεκτα, είναι η, δυναμική της εξέλιξης του ευρωπαϊκού δικαίου. Εάν κάποιο λοιπόν χρησιμοποιεί αυτές τι εξελίξεις θα πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα διάφορα παρακλάδια και όταν αναφερόμαστε σε κοινέ ή ελάχιστες προδιαγραφέ, θα πρέπει να σκεφτούμε ε, τι συνέπειες έχουν αυτά σε κάθε παρακλάδι. Υπάρχουν λοιπόν συνέπειες που μπορεί να έχει το ένα στο άλλο και σε κάποιο βαθμό υπάρχουν ήδη αυτές οι συνέπειες. Όταν συζητούμε λοιπόν κοινέ προδιαγραφέ, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά τη σταγματική νομοθετική εντολή που ίσως περιορίζει τις επιλογές που έχουν οι νομοθέτες. Σαφώς και υπάρχει το θέμα της νομικής βάσης. Ο περιορισμός του διασυνοριακού στο άρθρο 21 και ε, για μέτρα τα οποία σχετίζονται με κάθε τομέα περιορίζονται για κάθε συγκεκριμένο τομέα και μόνο. Παραδείγματο χάρη θέματα καταναλωτή, ανταγωνισμού και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και ο περιορισμός του άρθρου 114, το περιορισμός της εσωτερική αγοράς. Τα μέλη της Επιτροπής σας γνωρίζουν αυτό, που έχουμε, ε, αυτό το οποίο αποτελώ ε, το απογορευμένο ζήτημα της επικουρικότητας ε, το οποίο πλέον είναι μια πολιτική πραγματικότητα και μια συζήτηση στην Ευρώπη για το πόσο θα πρέπει να προχωρήσει το θέμα αυτό και τι θα πρέπει να γίνει με τις νομικές διαδικασίες. Στο θέμα των διαβουλεύσεων για τις αποσημειώσεις, ε, διαπιστώσαμε ότι πολλά κράτη-μέλη όταν απάντησαν στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αρκετά επιφυλακτικοί για το πόσο θα πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη. Εμείς το γνωρίζουμε ε, και το αποκαλούμε συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ότι θα πρέπει να εκχωρήσουν περισσότερα και πολλοί αναφέρονται και στη σημασία ε, επιτευγμάτων και σε επίπεδο κράτους μέλους, γιατί έχουμε εξελίξεις και εκεί. Και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς στην Ευρώπη, σε υπερεθνικό επίπεδο, θα έπρεπε τουλάχιστον σε κάποια μορφή διαλόγου να εντάσσεται και στην εθνική συζήτηση και στις εξελίξεις. Και επίσης έχουμε αυτό που ανέφερε και ο καθηγητής ε, ε, τις διάφορες ε, πολιτικές υφέρπουσες ιδέες της ε, εσωτερικής αγοράς, της ασφάλειας και της δικαιοσύνη. Ποιον βοηθάμε, τους καταναλωτές, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους πιστωτές ή τις οικογένειες. Βεβαίως αυτό αποτελεί επιλογή πολιτική. Ποιον θέλουμε να βοηθήσουμε και γιατί. Αυτό θα πρέπει να το επιλέξουν πολιτική. Και βεβαίως εδώ έρχεται να προσθεθεί και η συζήτηση ε, του πόσο ολοκλήρωση επιθυμούμε. Ε, σε δικονομικό επίπεδο ε, έχουμε το θέμα της αμαβαίας αναγνώρισης. Το να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε διαδικαστικές κανόνες ή αμοιβέ προδιαγραφές, κυρίως υπό την αιγίδα του άρθρου 21, στη Συνθήκη τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα σημαντικό ε, στοιχείο που μας αποσχολεί, αλλά ίσως αυτό το οποίο μας διέφυγε είναι ότι η αμοιβαία αναγνώριση δεν αποτελούσε ποτέ το επίκεντρο και ποτέ δεν ήταν ε, ξεκάθαρη ε, και ίσως θα θυμάστε και από την υπόθεση του Κασίς Δεντιζόν ε, προήλθε από διάφορα σημεία εξαιρέσεων και προστασίας των εθνικών προτύπων και προστασίας των ελαχίστων δικαιωμάτων στην ουσία. Όταν λοιπόν υπερβαίνουμε τα όρια της αμοιβαίας αναγνώρισης ε, στην ποινική δικαιοσύνη, Κάποιοι προσπαθούν να πούν ότι η αμοιβή εμπιστοσύνη θα ρυθμίσει όλα τα δυνητικά προβλήματα της αμοιβαίας αναγνώρισης ε, χωρίς δικλείδες ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί. Αλλά το θέμα είναι αν μπορούμε να επιβάλλουμε εκ των άνω αμοιβαία εμπιστοσύνη. Είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί ακόμα στην Ευρώπη και εγώ θα μπορούσα να πω ότι δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε εκ των άνω. Δεν μπορεί να την επιβάλλουν οι πολιτικοί την αμοιβαία εμπιστοσύνη χωρί να υπάρχει μια δυνατότητα ρύθμιση και στα δικαστήρια και στου ανθρώπου που ασκούν νομικά ε, επαγγέλματα και στην ε, δικαιοσύνη σε τοπικό επίπεδο. Πού μας οδηγεί αυτό λοιπόν. Υπάρχει αρκετή αμοιβή αναγνώριση στα διάφορα μέτρα στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους διάφορους κανονισμούς ε, ε, ε, στον κανονισμό για τις μικρές απαιτήσει, για παράδειγμα υπάρχουν κάποια στοιχεία αμοιβή αναγνώρισης. Το θέμα είναι αν χρειαζόμαστε περισσότερο, χρειαζόμαστε κάποιε κοινέ προδιαγραφέ ή υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσουμε τι πιέσει αυτέ και τα προβλήματα που προκύπτουν. Όπως ε, είπε και ο καθηγητές ε, Χες, αλλά όπως ε, έχει πει και η κυρία Γουόλης που κάθεται από την άλλη πλευρά, οι κοινέ προδιαγραφές μπορεί να είναι μια χρήσιμη λύση και ένα χρήσιμο πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουμε και κάποια από τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει με την αμοιβαία αναγνώριση χωρίς σε κάποιες περιπτώσει δικλείδε ασφαλεία. Προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα. Ποια κοινά πρότυπα ή του είδους κοινά πρότυπα θέλουμε. Θέλουμε ελάχιστα πρότυπα ή μέγιστα τέτοια πρότυπα. Θα αναζητήσουμε τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, θα αναζητήσουμε λεπτομερέστατα τέτοια πρότυπα πολιτικής δικονομίας. Πρέπει ακόμα τα ζητήματα αυτά που εκκρεμούν να τα επιλύσουμε. Και όπως είπε ο καθηγητής Χες πριν από λίγο, ως προς αυτό η, η εφιστάμενη μελέτη που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Νομικής μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε αν μπορούμε τελικά να καταλήξουμε σε κάποιο μοντέλο, σε κάποια ευρωπαϊκά ελάχιστα πρότυπα. Και αυτό, ξέρετε, αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί πολύ συχνά σταματάμε απλώς σε μια συγκριτική αξιολόγηση. Κάνουμε μια έρευνα συγκριτικής αξιολόγησης, βλέπουμε πού διαφέρουν τα συστήματα στην Ευρώπη, χωρίς όμως να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα. Το σχέδιο λοιπόν αυτό, η έρευνα αυτή βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κάποια ελάχιστα πρότυπα, σε έναν ελάχιστο κοινό παρανομαστή, επί του οποίου θα μπορούσαμε όλοι να συμφωνήσουμε, χωρίς όμως να θέλουμε να μπούμε πάρα πολύ στην αρμοδιότητα των εθνικών κρατών μελών της εθνικής δικαιοδοσίας. Ανταυτού νομίζω ότι η πιο εύστοχη πρακτική θα ήταν να ερευνήσουμε περισσότερο τα συστήματα εθνικής δικαιοδοσίας και εκεί πέρα να καταφέρουμε να καταλήξουμε στο καλύτερο εθνικό μοντέλο και αυτό να αποτελέσει επί τα αντικείμενο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Δεν έχουμε όμως φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Πρωτού ολοκληρώσω την παρουσίαση αυτή, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε από ποιο επίπεδο θα πρέπει να ξεκινήσουμε και ποιοι θα πρέπει να είναι οι πρώτοι παράγοντες οι οποίοι θα εμπλακούν. Ας μην είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα επιβάλλουμε εκ των άνω. Ας μην θεωρήσουμε ότι αυτή είναι εργασία μόνο ενό ανώτατου ρυθμιστή, ο οποίος θα πρέπει να επιβάλλει κοινά πρότυπα για όλη την Ευρώπη οι ίδιοι δικαστέ, οι ίδιοι επαγγελματίε του νομικού τομέα, οι νομομαθεί και δικηγόροι θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Και ορισμένοι για πρώτη φορά ασχολούνται πλέον με τον κανονισμό αυτών των μικρών, των προσφυγών ίσονο σημασία. Και Μόνο πρόσφατα άρχισαν κάποιοι νομομαθείς να ασχολούνται και να εφαρμόζουν αυτή τη νέα κοινοτική νομοθεσία. Δεν μπορούν όλα να γίνουν λοιπόν με μία νυχτή. Βρισκόμαστε προφανώς στην αρχή του εγχειρήματο αυτού, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε με ένα μαγικό ραβδί να αλλάξουμε τα πάντα από τη μία στιγμή στην άλλη. Θα απαιτηθεί χρόνος προκειμένου να δούμε πώς θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό επίπεδο προτύπων, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Πάντω αυτό που είναι το πιο σημαντικό και αυτό που, και αυτό που με κάνει αισιόδοξη είναι το ότι ήδη έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και είμαστε όλοι έτοιμοι να αρχίσουμε να κάνουμε μία συζήτηση για την καλύτερη δυνατή στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε ένα, σενάριο το οποίο όπως όλοι είδατε είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και πολύ σχηδές. Σας ε, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ε, κυρία Εύα Στορτπρουκ από το Πανεπιστήμιο της Σουψάλα και τώρα μπορεί να ξεκινήσει και η συζήτηση. Και προφανώς όμως ε, θα θέλαμε να ακούσουμε και την Ταϊάννα Γόλης αλλά και τον κύριο Σότερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε πάντως το λόγο. Νταϊάννα, θέλετε μήπως εσείς να πάρετε πρώτο το λόγο. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκλησή σας Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ακούσω την παρουσίαση του κυρίου Χές, καθώς επίσης και την παρουσίαση της κυρίας Στόρσκμπρουκ. Ξέρετε ότι ε, και από την ε, πρώτη εργασία που έχω κάνει εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από την υφιστάμενη θέση που έχω στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Νομικής, ασχολούμαι με τα ζητήματα αυτά. Να αναφερθώ σε τρεις θεματικές ενότητες ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να γνωρίζετε. Χρησιμότητα, συνέπεια και τεχνολογία. Αυτά είναι τα τρία θέματα τα οποία κρίνουν ιδιαίτερα σημαντικά. Πρώτον, συνεκτικότητα, συνέπεια, ζήτημα το οποίο έθιξαν και προαλήσαντες. Είναι πάντως σαφές ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα αποκλίνουν από τη μία χώρα στην άλλη, οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές. Από τη μία πλευρά αυτό εμπλουτίζει την όλη συζήτηση, μα δίνει πολλές διαφορετικές συναλλακτικέ, από την άλλη όμως ενδεχομένω αυτό να περιπλέκει και κάπως τα πράγματα. Να είναι δύσκολο δηλαδή να καταλήξουμε σε μια κοινή εικόνα και προκύπτουν και κάποια νέα προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η συνέπεια, η συνεκτικότητα να διέπει οποιαδήποτε μελλοντική μα νομοθεσία. Να αναφερθώ τώρα και στο ζήτημα της χρησιμότητος. Δηλαδή, για ποιο λόγο θα πρέπει εμείς και αναφέρομαι στον πρώτο πρόσωπο του να προχωρήσουμε με το εγχείρημα αυτό. Γιατί προφανώς μιλάμε αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους πολίτες και ουσιαστικά απότερος στόχος μας είναι να απλοποιήσουμε τη ζωή των πολιτών και να έχουν πιο εύκολη και ομαλή πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Νομικής ως κοινότητα δικηγόρων προσεγγίζουμε το ζήτημα αυτό. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να, αναφερθούμε, να εμπλέξουμε δικαστές, δικηγόρους οι οποίοι διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, αλλά και δικηγόρους οι οποίοι ασκούν στην πράξη στο επάγγελμα. Και όλοι αυτοί οι χρήστες ε, της πολιτικής δικονομίας ουσιαστικά μας λένε ότι κάτι δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή πολύ καλά. Θέλουμε λοιπόν να καταστήσουμε το σύστημα πολιτικής δικονομίας πιο λειτουργικό να είναι σε θέση άμεσα να λειτουργήσει και να ελοποιηθεί. Ας μην διστάζουμε λοιπόν και ας μην λέμε ότι το εγχείρημα αυτό μπορεί να αποτελέσει απειλή για τα κράτη-μέλη. Δεν θα είναι απειλή αν είναι σε θέση να δώσει στα κράτη-μέλη κάτι το οποίο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τους πολίτες, από τους επαγγελματίες του τομέα της νομικής, κάτι το οποίο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της εσωτερικής αγοράς. Αλλά χρειαζόμαστε ένα σύστημα πολιτικής δικονομίας το οποίο θα είναι προσβάσιμο συνεκτικό παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος να αφαιρθώ στην τεχνολογία. Αναφερθήκαμε πριν από λίγο στις νέες τεχνολογίες που ενδεχομένω να παρακολύουν την παροχή της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μολονότι όμως μπορεί να δημιουργούν κάποια προβλήματα, από την άλλη μπορεί να διευκολύνουν και την ε, απονομή της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι ε, Απομένει να δούμε με πρωτοβουλία του Συμβουλίου πώς μπορεί να βελτιωθεί το Portal e-Justice, αυτή η ηλεκτρονική πύλη δικαιοσύνης. Πρέπει να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που έχουμε στο διαδίκτυο, να δούμε πώς μπορούν όλες αυτές τις πληροφορίες να μας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις ευρωπαϊκές διατάξεις που ήδη υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για αυτές τις προσφυγές ίσονος σημασίας. Επίσης, μέσω της τεχνολογίας θα είμαστε σε θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχουμε και ένα σύστημα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών. Προκειμένου όμως να γίνουν όλα αυτά και προκειμένου όλα αυτά να αποτελούν συνεκτικά μέρη ενός ενιαίου συστήματος, θα πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός, ορισμένα πράγματα λειτουργούν σε κάποιους τομείς και μερικώς μόνο. Χρειαζόμαστε λοιπόν να προσδώσουμε στο σύστημα μεγαλύτερη συνεκτικότητα και διαφάνεια και κατά αυτόν τον τρόπο ελπίζω ότι θα καταφέρουμε πραγματικά να δώσουμε στους πολίτες καλύτερη και πιο εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ζήτημα το οποίο όπως γνωρίζετε μας είχε απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας ευχαριστούμε. Ακούσαμε την Ταϊάννα Γόλη, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Νομικού Ινστιτούτου. Ο κύριος Μπούντα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε ένα ζήτημα το οποίο μας προκαλεί κάποιες ανησυχίες, γιατί σε τελευταία ανάλυση όλοι μας συμμετέχουμε ενεργώς στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και όλοι μας θέλουμε μία δωρεάν, εύκολη, γρήγορη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες. Αυτός είναι ο απότερος στόχος μας. Δυστυχώς όμως Οφείλω να πω, και το λέω αυτό διότι είμαι σκιώδης εισηγητής για την διαδικασία small claims, ότι πολλά κράτη-μέλη είναι ιδιαίτερα διστακτικά όσον αφορά τα ελάχιστα αυτά πρότυπα πολιτικής δικονομίας. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν είναι ότι τα κράτη-μέλη με τη δράση τους δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσαμε όλοι να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σιγά σιγά μέσω παραχωρήσεων από όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργηθούν τα απαραίτητα μέσα που θα οδηγήσουν σε μια κοινή πολιτική δικονομία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο διστάζουν τόσο πολύ τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι όλες αυτές οι νέες διαδικασίες εξυπηρετούν ουσιαστικά τον ίδιο τον πολίτη αλλά και το ίδιο το κράτος μέλος και εξυπηρετούν επίση και τα συμφέροντα των ίδιων των επιχειρήσεων μας τέθη το ερώτημα ποιον ακριβώς εκπροσωπείτε. Μα δεν εκπροσωπούμε ούτε μεμονωμένα τους πολίτες, ούτε μεμονωμένες επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε κατά τρόπο ισορροπημένο και αντικειμενικό τους πάντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν μεροληπτήσουμε, αν τεθούμε με τη μία ή την άλλη πλευρά, με τους πολίτες ή με τις επιχειρήσεις, το σύστημα προφανώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Ξέρετε ότι ε, όλοι κινούμεθα στα πλαίσια ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου Ξέρετε ότι έχουμε νομοθετήσει πάρα πολύ στο παρελθόν, έχουμε όλες αυτές τις συνθήκες, έχουμε τα νομοθετήματα Βρυξέλλες 1 και Βρυξέλλες 2 και όλα αυτά τα έγγραφα βασικά δεν μπορούν να γίνουν ποτέ πραγματικότητα αν δεν υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση. Να αναφερθώ για παράδειγμα σε μια δικαστική διαφορά που μπορεί να προκύψει στην εργασιακή νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών. Μέσω της νομοθεσίας Βρυξέλλες 1, ένας εργαζόμενος ο οποίος εργάζεται εκτός της χώρας πρόλευσής του δεν μπορεί να στραφεί κατά του εργοτότη του στη χώρα υποδοχής. Προβλέπεται ότι μπορεί μόνο στη χώρα προελευσής του, στη χώρα καταγωγής του να κάνει μια τέτοια προσφυγή. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο πρέπει να μπορεί ο πολίτης αυτός, ο οποίος προέρχεται από μια άλλη χώρα, να μπορεί να στραφεί κατά του εργοδότη του και στη χώρα υποδοχή, στη χώρα στην οποία ουσιαστικά εργάζεται. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις παρουσιάσεις που κάνατε, γιατί πραγματικά καταδεικνύουν ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να καταστήσουμε τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Mr. Schotter would Ευχαριστώ. Κύριε Σότερ, θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι πρόκειται πράγματα για ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό ζήτημα. Τα δικαιονομικά δικαιώματα έχουν μεγάλη σημασία και όχι μόνο στο δικαστικό τομέα στον οποίο έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος αλλά και σε επίπεδο αστικής δικαιοσύνη όπου τα πράγματα έχουν εξελιχθεί με λίγο διαφορετικό τρόπο και ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές παρουσιάσεις από τους ε, παρακαθήμενους για το πόσο ε, ζωφερή είναι η εικόνα και πώς ε, αναπτύχθηκε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Ακούσαμε τώρα τον κύριο Μπούντα να αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό μέσο, το οποίο αυτή τη στιγμή αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά τα διαφορετικά μέσα τρόπον την να έχουν ε, ασχοληθεί με τα δικονομικά δικαιώματα και πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό τα αποτελέσματα ε, ήταν ποικίλα. Αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτό είναι κάτι καλό ή κάτι κακό. Τελικώ νομίζω ότι θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό με την Diana Wallis. Πρέπει να είναι στόχος μας ε, να υπάρξει συνοχή και να κινηθούμε προς τη συνοχή. θα αναφερθώ σε ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2014, το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δικαιοσύνης για το 2020 και ε, εξετάζει μια διαδικασία για τη δικαιοσύνη και έφτασε ε, το μεγάλο ερωτηματικό προς τα πού θα πρέπει να κατευθυνθούμε για τα επόμενα χρόνια. Και ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία αυτού του εγγράφου ήταν το γεγονός ότι θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς ε, μεγαλύτερη κωδικοποίηση, μεγαλύτερη συνοχή. Σίγουρα αυτό αποτελεί στοιχείο της διαδικασίας. Ο στόχος αυτός όμως, παρά το γεγονός ότι είναι αξιοζήλευτος, θα πρέπει να ίσως τα σκελιστεί και με πολλούς άλλους στόχους, ε, ώστε να υπάρξει πρόοδος για να υπάρχει ολοκλήρωση του κεκτημένου μας με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε. Ορισμένες φορές ε, μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία, ορισμένες φορές ε, πρέπει να κινηθούμε ε, με μεγαλύτερη φιλοδοξία, με, λιγότερη φιλοδοξία από όσοι είχαμε αρχικά προβλέψει, αλλά το θέμα είναι η κατεύθυνση και κατά πόσον υπάρχει πρόοδος. Η διαδικασία, για παράδειγμα, για τις προσφυγές είναι σημασία. Να τη χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα. Είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία. Ε, δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες, αλλά είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία η οποία περιλαμβάνει πολλές καινοτομίε και περιλαμβάνει αυτή την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να συνδεθεί και με όλα τα εθνικά συστήματα και αυτό κάνει. Και φυσικά είναι μια διαδικασία να εξελίξει. έγινε μια αναθεώρηση και αυτή τη στιγμή ε, αναθεωρούμε ε, την νομοθεσία και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ χρήσιμες βελτιώσεις στην όλη διαδικασία για τις προσφυγές αυτές. Ε, αλλά σίγουρα θα υπάρξει και μία εξέταση αργότερα. Θα είναι μια διαδικασία η οποία θα προχωρήσει βαθμιδών. Και νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να πω ότι δεν περιορίζεται στην ευρωπαϊκή διαδικασία για τις προσφυγές ίσονος σημασίας. Ε, κάνουμε και μια αξιολόγηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α στον τομέα οικογενειακού δικαίου, που είναι πάλι ένας πολύ σημαντικός τομέας. Και επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα των ελαχίστων προδιαγραφών και το εξετάζουμε αυτό το θέμα. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει τώρα να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά με οριζόντιο τρόπο. Αν θα είναι αυτό κάτι καλό ή αν θα μας ε, παρακολύσει αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και πολύ συγκεκριμένα και χρήσιμα βήματα προς την κατεύθυνση που εξετάζουμε για κάθε μεμονωμένο νομοθέτημα. Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάστηκε να το αξιολύσουμε αυτό στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ελοκλήρωσης. Είναι το αρχαίο δίλημα του πώς προχωράει κανείς. Ε, τελικώς νομίζω ότι θα βρούμε έναν τρόπο ο οποίος ε, θα είναι χρήσιμος, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ε, προχωρούμε πάντα. Ήθελα επίσης να αναφέρω και τις άλλες ε, πτυχές που ανέφερε η κυρία Στόρς Κρόπ και θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Υπάρχει ε, αυτό το ο πίνακα επιδόσεων δικαιοσύνη, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, το e-justice και επίση θα ήθελα να σταθώ και σε δίκτυα όπω το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. Όλα αυτά τα εργαλεία αποτελούν μέσα ε, βάσει των οποίων δημιουργείται ε, μια κοινή κουλτούρα της ε, συνεργασίας μεταξύ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επίσης ε, της όλης εθνικής διαδικασίας επί των οποίων βασίζονται αυτές οι διαδικασίες. Είναι μια ε, συνεχώς ε, εναλλασσόμενη διαδικασία και φυσικά υπάρχει και όλη αυτή η χρήσιμη ε, διαδικασία που γίνεται και ε, χαίρεται που την παρακολουθεί ως παρατηρητής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είμαι βέβαιος ότι θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα μας οδηγήσουν στη συγκεκριμένη αλλαγή νοοτροπίας. Ε, χαίρομαι ε, που γίνεται αυτή η συζήτηση και με τα χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριος Ράνιεφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να έχουμε μια πιο διαρθρωμένη, μια πιο συνεκτική προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πολιτική δικονομία των κρατών μελών. Τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο η ανάγκη να έχουμε κάποια ευρωπαϊκά ελάχιστα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες κοινέ προδιαγραφές όσον αφορά την πολιτική δικονομία, προκειμένου να μπορούν να αναγνωρίζονται παντού οι αποφάσεις δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουμε να έχουμε απόλυτη αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών εθνικών αποφάσεων. Θα πρέπει να κατοχυρώνονται τα πολιτικά, τα δικαιώματα πολιτικής δικονομίας όλων των Ευρωπαίων πολιτών παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα της δικαιοδοσίας που επεμβαίνει στα πλαίσια μιας δίκης. Η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών αυτών ελάχιστων προτύπων στην εθνική πολιτική δικονομία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομεί όπου θα πρέπει να γίνουν περισσότερε αλλαγέ προκειμένου να καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ότι θα πρέπει να γίνει απαραίτητη κωδικοποίηση για λόγου νομική ασφάλεια. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ποια μέθοδο θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Εγώ προτείνω μέσα τα οποία θα πρέπει να είναι κοινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι σε ορισμένε περιπτώσει, ιδίω με την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό μέσο ή, για παράδειγμα, μέσω του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Ασύλληψη. Ξέρετε ότι έχουμε καταφέρει στα πλαίσια αυτών των ευρωπαϊκών διαδικασιών να εξασφαλίσουμε μια οριζόντια εφαρμογή κάποιων δικαιωμάτων. Αυτό έχει γίνει επίση και για την προστασία των καταναλωτών αλλά και για το δίκαιο ανταγωνισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, πολύ σύντομα. Την εισήγηση του καθηγητού Θέσα από την οποία έχω χάσει σημαντικά στοιχεία και έτσι κατά το μάλλον ήταν μόνο το τελικό τμήμα των συμπερασμάτων της ε, κυρίας προλαλήσάς σας ε, άκουσα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά γιατί είναι τόσο ενδιαφέρον να μπορεί κανείς να παρακολουθεί αυτά. Αναφέρατε αν λειτουργούν αυτά και αν θα μπορεί κανείς να επιβάλλει την εμπιστοσύνη εκ των άνω προς τα κάτω και με την αναγκαία αμοιβαιότητα αναγνώρισης, με την ε, αμοιβαία αναγνώριση πρέπει να προχωρήσουμε σε εκείνους τους τομείς όπου δεν είναι δυνατόν να έχουμε την ομοφωνία στο Συμβούλιο. Και έτσι με πάρα πολύ επικοδομητικές συναντήσεις καταλήξαμε σε μια πολύ θετική συνεργασία που υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ε, με μεγάλη εξειδίκευση και με βάση την ομολογία του 10 μπορούμε να προχωρήσουμε. Ακόμα και αν με ντεμίνιμις, με ελάχιστες ε, προδιαγραφές, ε, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει μία παρεκκλίνουσα διαδικασία. Θα ήθελα να αναφέρω αυτό. Ακριβώς εμείς σε αυτή την αίθουσα για την προστασία, την νομική προστασία μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και να μπορέσουμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Δηλαδή ένα έργο που ιδιαίτερα κατά την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία από πλευράς Μπερλιγκουέρη είχε προαχθεί για την καλύτερη συνεργασία βέλτιστη συνεργασία για την επιμόρφωση και περαιτέρω κατάρτιση των δικαστών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σχέση με τους στόχους που εσείς ε, αναφέρατε, ώστε να υπάρξει μια κοινή μέθοδος ε, όπου είναι αναγκαίο σε κάποιους τομείς να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ε, και τις προκλήσεις. Πολλοί πολίτες λένε αφενός ότι υπάρχει η εθνική ρύθμιση και έχουμε από την άλλη πλευρά ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν όπως για παράδειγμα για το οικογενειακό δίκαιο όταν για ένα διαζύγιο ή όταν περιουσιακά στοιχεία αμφισβητούνται ή διεκδικούνται να μπορούν να, τα θέματα αυτά να προαθούν χάρη των πολιτών. Είμαι πεπισμένη ότι τα αστικά θέματα δεν θα πρέπει ε, ιδεολογικά να διαμορφώνονται, θα πρέπει καλύτερα να μπορέσουν να προαθούν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να δούμε πώς μπορεί να γίνει με τη βελτίωση των προδιαγραφών, με την αμοιβαία αναγνώριση προδιαγραφών και διαδικασιών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εμείς από πλευράς ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ζητήσουμε να υπάρξει μεγαλύτερη ακρίβεια και ακριβολογία ώστε πριν υπάρξει μια τελική ρύθμιση να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε τα πλαίσια. Όπως είπα, μόνο τα τελευταία στοιχεία της εισήγησης μπόρεσα να ακούσω. Έχασα την το προηγούμενο μέρος της παρέμβασης. Ευχαριστώ. Ε, Η κυρία Ντελβό, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές θεωρώ ότι αποτελούν έμπνευση και είναι πολύ επικοδομητικές οι παρουσιάσεις. Με πάσα ταπεινοφροσύνη λοιπόν, εγώ πρέπει να πω ότι εγώ ανακαλύπτω τις όλες διαδικασίες σε θέματα αστικού δικαίου. Στην αρχή είχα πει ότι είναι πάρα πολλά τα μέσα, πώς μπορεί ένας απλός πολίτης να γνωρίζει σε ποιον αποτανθεί, πώς ε, θα βρούμε νομικούς που θα γνωρίζουν όλες αυτές τις διαδικασίες στις χώρες τους, διότι ο καθηγητής ε, Χές αναφέρθηκε στο Λουξεμβούργο που ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για το ε, σύστημα της δικαιοσύνης του, αλλά δαπανούμε όλοι πολλά χρήματα για όλα αυτά. Αυτά δεν σημαίνει ότι αναλογικά η ποιότητα είναι αντίστοιχη της δαπάνης που γίνεται και πιστεύω ακόμα ότι και σε αυτές τις χώρες που δαπανώνται πολλά χρήματα δεν είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί ο νομικός ο οποίος θα σας καθοδηγήσει προς τη σωστή διαδικασία εάν δεν γνωρίζετε κι εσείς τα πράγματα εκ των έσω ε, στον τομέα. Εγώ θέλω όμως να παραμείνω αισιόδοξη και βεβαίως ε, σας ενθαρρύνω και υποστηρίζω ε, ακράδαντα την ε, συνέπεια θεωρώ ότι πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμα αυτά τα στοιχεία και θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια. Όμως δεν γνωρίζω ακριβώς και εδώ θα ήθελα να ε, μου πούνε οι ειδικοί πώς μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη συνοχή. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτή η διαδικασία των ελάχιστων προδιαγραφών ε, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί σχετικά αποτελεσματικά. Σαφώς και θα θέλαμε να υπάρχει μια κωδικοποίηση να μπορούν να γίνουν τα πάντα γιατί και θα ήταν καλό και θα είχαμε μια πλήρη εικόνα αλλά είμαι μάλλον επιφυλακτική μετά από τη μικρή εμπειρία που είχα διότι θεωρώ ότι αν θελήσουμε να έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό θα περιπλέξουμε πολύ τα πράγματα και δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και έχω και κάποιες ερωτήσεις για τη συνεργασία μεταξύ δικαστή και εμπειρογνωμένων σε κάθε χώρα. Υπάρχει ένα δίκτυο, υπάρχουν ε, ε, μαθήματα κατάρτισης και επιμόρφωσης και θα ήθελα να γνωρίζω ποιο ποσοστό των ε, ειδικών του δικαίου μπορούμε να βοηθήσουμε. Ε, έχουμε κάποια εικόνα για το πόσο χρόνο θα χρειαστεί, διότι η διαδικασία είναι μακρά, μεν, αλλά θα ήθελα να έχω και μια προοπτική της ε, τελικής ε, επιτυχίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος από τα μέλη το λόγο. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι λοιπόν θέλουν να σχολιάσουν αυτά τα οποία ακούστηκαν. Ο καθηγητής Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να δώσω συνέχεια και να αναφερθώ σε αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε. Αλλά μπορώ να μιλήσω γερμανικά, έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να αποσαφινιστεί ότι για τον μέσο δικαστή στην Ευρώπη ο αριθμός των διασυνοριακών υποθέσεων είναι περίπου 1 έως 5% και δεν έχουν πείρα ή βιώματα σχετικά. Και αν έχουμε ετερογενείς περιπτώσεις ε, και διατάξεις, κάθε φορά πρέπει από μηδενικού σημείου να ξεκινά κανείς και να μαθαίνει. Και αυτό είναι ιδιαίτερα δαπανηρό και για τους ε, δικηγόρους. Καλούνται τα κράτη-μέλη λοιπόν να δράσουν. Ο κανονισμός Μπαγκατέλη είναι ένα παράδειγμα λοιπόν κακής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη. Δεν είναι γνωστός λοιπόν ο κανονισμός αυτός. Στον κανονισμό θα πρέπει διατάξεις και ε, ρήτρε να εμπεριέχονται που θα υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να δημοσιοποιούν τα στοιχεία αυτά και να γνωστοποιούν τα στατιστικά στοιχεία ώστε να είναι περισσότερο ας το πω έτσι προσπελάσιμα ο κανονισμός είναι ένα καλό μέσο όμως δεν μπορεί να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται η οδηγία είναι πολύ καλύτερη γιατί στο τέλος τέλος τα θέματα εφαρμογής μπορούν να ελεγχθούν και να προαχθούν αυτό θα έπρεπε να το σκεφτούμε είναι ένα σημαντικό στοιχείο απλούστευση να μην έχουμε πολύ εξειδικευμένους κανονισμούς από την άλλη πλευρά όταν προτείνονται να καταργηθούν κάποια πράγματα, για παράδειγμα αναφέρθηκε για ένα κανονισμό ότι δεν το χρειαζόμαστε σε σχέση με αυτή την πτυχή πια. Όμως όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται οι κανονισμοί δεύτερης γενεάς, δηλαδή οι διατάξεις που εγκρίνονται μετά από αυτή την πρώτη ε, φάση θα έπρεπε τα κράτη-μέλη στα εθνικά πλαίσια τα δικονομικά να εντάξουν διατάξεις που θα αναφέρονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και αυτό θα μπορούσε να είναι δεσμευτικό μέσω της ευρωπαϊκής οδηγίας. Είμαι υπέρ μικρών βήματων. Μικρά βήματα πρέπει να κάνουμε, αλλά μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε και να δούμε πού βρίσκονται τα ουσιαστικά προβλήματα, αλλά και ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές τι λειτουργεί καλά και τι μπορούμε να ε, μάθουμε από αυτά. Έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Thank you σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μια-δυο παρατηρήσεις να κάνω. Πρώτον, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ότι μιλάμε για τα δίκτυα αυτά και για τους εθνικούς δικαστές και για το ρόλο που διδραματίζουν οι εθνικοί δικαστές στο λεγόμενο ευρωπαϊκό αρχιτεκτόνημα. Δεν θέλω να ακούγομαι σαν μια παροχημένη φωνή, αλλά όταν ήμουν εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαμε και μια έκθεση για το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι αξίζει να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα και να δούμε τι, τι πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την ε, γνώση και τη δέσμευση που έχουμε πλέον στον τομέα αυτό των εθνικών δικαστών. Σίγουρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, αλλά πολύ συχνά με πολύ αργό ρυθμό. Νομίζω ότι αναφερθήκατε και σε αυτό το ζήτημα της συνέπειας, της συνεκτικότητος. Ναι, μα προφανώς θα πρέπει να σημειωθεί η προόδος πολύ προσεκτικά, δείχνοντας την απαραίτητη ευαισθησία και πολλές φορές βέβαια ο ρυθμός που υιοθετούμε είναι ιδιαίτερα αργός. Αυτό που θα έλεγα όμως κυρίως είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε προς τα πού πηγαίνουμε, ποιος είναι ο τελικός μας προορισμός και πώς τελικά τα πράγματα θα έρθουν να δέσουν στο τέλος. Αυτό θα πρέπει να δούμε. Γιατί αν συνεχίσουμε με αυτόν τον μεμονωμένο, κατακαιρματισμένο τρόπο εργασίας, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό προορισμό. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι η εργασία που επιτελούμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Νομικής μπορεί όντως να βοηθήσει τα πράγματα, γιατί μπορεί πραγματικά να καταφέρνει να μας, να μας... Να μας βοηθήσει να καταλάβουμε, να δούμε πού πηγαίνουμε. Μολονότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε μέσω του Ινστιτούτου αυτού μία σφαιρική απάντηση, τουλάχιστον έχουμε κάποιους εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα έχουν ασχοληθεί με όλα τα κρεμή ζητήματα και θα μπορέσουν να δώσουν αν μη τι άλλο κάποιες απαντήσεις. Στα πλαίσια του Unit 1 έχουμε ένα οργανισμό ο οποίος βασίζεται στα κράτη-μέλη και αν σε τελική ανάλυση τα ίδια τα κράτη-μέλη επιθυμούν να προωθήσουν την εργασία αυτού του οργανισμού, τότε μέσω του οργανισμού αυτού πραγματικά θα δώσουν, πιστεύω, απαντήσει σε πολλά από τα ερωτήματα που ακούσαμε σήμερα. Ελπίζω να σας κάλυψα με την απάντηση αυτή. Ναι, και εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο θυμήθηκα μόλις ολοκλήρωσα την παρέμβασή μου πριν από λίγο. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ε, σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται ατενίζοντα το μέλλον και συμφωνώ απόλυτα με την Ταϊάννα Γόλη, προφανώ θα πρέπει να γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε, ποιο είναι ο προορισμό μα. Αυτό πιστεύω ότι θα μα καθοδηγήσει. Προφανώ θα πρέπει να κινούμεθα βαθμιδών, κοιτώντα κάθε φορά προ ποια κατεύθυνση αξίζει περισσότερο να κινηθούμε, αλλά κάθε φορά θα πρέπει να δούμε πώ εξυπηρετούμε τελικά τα συμφέροντα του πολίτη, τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Μπορεί τα πράγματα να φαίνονται κάπως αποσπασματικά, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε κάπου έναν οδικό χάρτη, αφού γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε, τότε νομίζω ότι η εργασία μας δεν μπορεί παρά να είναι ποιοτική. Και θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω σε ένα ζήτημα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό, το ζήτημα της καλύτερης νομοθεσίας. Η καλύτερη αυτή νομοθεσία, η βελτιωμένη νομοθεσία, μπορεί να αποτελέσει πραγματικά καθοδηγητή. Και θα πρέπει πάντα να αξιολογούμε και τις επιπτώσεις της νομοθεσίας. Προφανώς θα πρέπει η πολιτική δικονομία της κάθε χώρας να γίνεται σεβαστή, αυτό μας λένε άλλωστε και συνθήκες, αλλά μην ξεχνάμε και ποιος είναι ο στόχος μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεχομένως να υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι επέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό μέσω μιας βελτιωμένης νομοθεσίας και μέσω μιας καλής κατανόησης του τι τελικά κάνουμε και πρέπει να σας πω ότι μόλις ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου ένα πρόγραμμα υποβολής προσφορών, ένα πρόγραμμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακριβώς για αυτό το ζήτημα της πολιτικής δικονομίας και επικεντρωνόμαστε σε δύο πολύ συγκεκριμένου τομείς της πολιτικής δικονομίας. Πριν από λίγο αναφερθήκαμε στο ότι θα πρέπει να καταργηθεί το εξκουατόρ, και η αναγνώριση της, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και μέσω λοιπόν μιας δικής μας μελέτης θέλουμε να δούμε πού έγκυται το πρόβλημα, πού βρίσκονται δυσκολίες, πού και πώς τροχοπεδετείται το όλο ζήτημα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, γιατί μόσο των συγκεκριμένων αυτών στοιχείων θα δούμε πού αξίζει να λάβουμε δράση. Είναι πολύ καλύτερο να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο από το να λέμε ότι θα πρέπει εκ των άνω να επιβάλλουμε ένα νέο σύστημα. Έτσι λοιπόν στις 2 Ιουνίου υποβλήθηκε αυτή η πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα εκπονηθεί μια μελέτη που νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και να αναφερθώ και στο δεύτερο ζήτημα, το ζήτημα της νομολογίας, της νομολογίας του δικαστηρίου όσον αφορά τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε ποια συμπεράσματα θα καταλήξουμε μέσω αυτής της νομολογίας του δικαστηρίου. Η όλη αυτή μελέτη θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι πολλοί θα ανταποκριθούν σε αυτή την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο. Πρέπει όμω να σα πω ακόμα ότι έχουμε στη διάθεσή μα κάποια πολύ σημαντικά μέσα όσον αφορά την πολιτική δικονομία. Τον κανονισμό, για παράδειγμα, για τι υπηρεσίε. Στα πλαίσια τη αναθεώρηση αυτού του κανονισμού, στα τέλη του 2013 καταλήξαμε σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα και ξεκινήσαμε και μία μελέτη προκειμένου να έχουμε μια πιο συγκριτική εικόνα των κανόνων που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά την πολιτική δικονομία. Νομίζω ότι εξετάζοντας μόνο την ομολογία και την πολιτική δικονομία των κρατών μελών μπορούμε να δούμε τελικά σε ποια επίπεδα υπάρχει συνεργασία και ποια ζητήματα ακόμα εκκρεμούν. Όσον αφορά τώρα το δίκτυο και όσον αφορά την κατάρτιση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα πάντα έχουν να κάνουν με την εφαρμογή και η εφαρμογή είναι πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε εμπορικά ζητήματα και αστικά, δική, αστικά ζητήματα. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός και επιτρέπει τελικά στους εμπειρογνώμονες και όχι μόνο στους δικαστές αλλά γενικότερα στους επαγγελματίες του τομέα και τους υπόλοιπους εμπλεκομένους να γνωρίζουν περισσότερο τι συμβαίνει όσον αφορά τα εθνικά συστήματα πολιτικής δικονομίας. και πραγματικά επαφιόμεθα πάρα πολύ στους εθνικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμμετέχουν στα δίκτυα αυτά προκειμένου να τα προβάλλουν περισσότερο. Θέλουμε κι εμείς να προωθήσουμε τα δίκτυα αυτά γιατί δυστυχώς δεν είναι παρκώς γνωστά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα και θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται περισσότερο. Για παράδειγμα η πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, το e-justice, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα προγράμματα κατάρτισης επίσης. Έχουμε θέσει ως στόχο να εκπαιδεύουμε, να καταρτίζουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό επαγγελματιών του νομικού τομέα. Η στρατηγική μας λοιπόν να καταφέρουμε να επηρεάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επαγγελματίες. Ο καθηγητής σχέση αναφέρθηκε επίσης στα στατιστικά δεδομένα. Δεν μπορεί κανείς να κάνει μία αξιόπιστη αξιολόγηση αν δεν χρησιμοποιεί στατιστικά δεδομένα. Και αυτό λοιπόν το αναλύουμε περισσότερο. Καταλαβαίνετε όμως ότι η συγκέντρωση και η συλλογή στατιστικών δεδομένων προποθέτει την ύπαρξη πόρων και οι πόροι συνήθως προέρχονται από τα Εθνικά Υπουργεία Δικαιοσύνης, από τα Εθνικά Συμβούλια Δικαιοσύνης. Ξέρετε όμως ότι αυτή τη στιγμή κινούμεθα σε μια συγκυρία οικονομική η οποία δεν μας επιτρέπει να έχουμε τους απαραίτητους πόρους. Πάντως, όταν κληθούμε να αναθεωρήσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να έχουμε κατά νου το γεγονός ότι χρειαζόμαστε ποσοτικοποιημένα στατιστικά στοιχεία προκειμένου πραγματικά να αξιολογούμε αξιόπιστα την κατάσταση κάθε φορά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ για αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα διάλογο, τα σχόλια, τις ερωτήσεις και είναι μια έμπνευση και ενθάρρυνση, προτροπή για μας που εργαζόμαστε σε αυτόν τον τομέα. Επί αρκετά χρόνια σε τρεις διαφορετικές νομολογίες εργάστηκα στην Ευρώπη και είδα ότι υπάρχουν και δικαστές που δεν έχουν κάποια ιδέα για, αυτές, για αυτή τη ρύθμιση και δεν μπορούν να την εφαρμόσουν και έτσι δημιουργείται ας το πω έτσι ένα πρόβλημα και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν και ελπίζουμε και στην κατάρτιση και εκπαίδευση νομική των εμπλεκόμενων και έτσι θα πρέπει να είναι επικοδομητικές αυτές οι διαδικασίες και είναι κάτι που προσπαθώ να προωθήσω και με το αξίωμα που έχω τώρα πολυσχηδή πράγματα πρέπει να γίνουν και είναι ενθαρρυντικά το ότι τα διαφορετικά ιδρύματα και θεσμοί εμπλέκονται στην ευρύτερη εικόνα για να ε, μπορέσει να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα σε αυτό το μείγμα που είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο Ευρωβουλευτή να ζητεί τον λόγο. Τότε ευχαριστώ για άλλη μία φορά τους ε, εξέχοντες προσκεκλημένους όσοι ε, συγητές που εξεφώνησαν τους λόγους τους ε, και μας εμπλούτησαν. Ο κύριος Χέσε έπρεπε να αποχωρήσει ήδη. Στους τρεις που απομένουν μπορούμε να τους αποχαιρετήσουμε. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που μας παρουσιάσατε τα βιώματα και τις γνώσεις σας και προσβλέπουμε στο να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Η σημερινή συζήτηση έδειξε ότι διεξάγεται σε μια αναγκαία χρονική στιγμή και, ήταν, και είναι αναγκαία. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το σημείο 6. Τροποποιήσεις, τροπολογίες στην επέκταση της προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μη γεωργικά προϊόντα. Και θα λάβει τον λόγο η εισηγήτρια κυρία Ροζιέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους μου για τις ε, τροπολογίες τους που δείχνουν λες και χρειαζόταν ότι υπάρχει συνένεση ε, ως προς ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τον επικοδομητικό χαρακτήρα των προτάσεών σας, διότι υπενθυμίζουν ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ευρωπαϊκή προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και για να διατηρηθεί η απασχόληση σε τοπικό επίπεδο και για να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις, κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις επιτόπου και φυσικά για τη βελτίωση σε θέματα τουριστικής προσέλκυσης ε, στη συγκεκριμένη περιοχή και φυσικά κατάλληλη ε, δυνατότητα για τους καταναλωτές να μπορούν να διαβάσουν την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν και αυτή την εγγύηση ότι η ε, προέλευση αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή και επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν επί τόπου και που έχουν τεχνογνωσία και μεθόδους παραγωγής σαφώς ε, καθορισμένες και ποιοτικέ. Επειδή πρόκειται για μια διάταξη η οποία απευθύνεται πρωτίστως ε, σε μικρές επιχειρήσεις, μπορεί και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, κάτι το οποίο επισημαίνεται από πολλούς ε, συναδέλφους της τροπολογίας και συμφωνώ κι εγώ απολύτως. Ε, θα πρέπει να είναι απλές οι διατάξεις και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φροντίσουμε και επίσης αυτές οι διατάξεις δεν θα πρέπει να αποτελούν πρόσκομα στην καινοτομία. Ε, να βοηθήσουν αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες ναι μεν ε, τηρούν την παράδοση αλλά μπορεί να αποτελέσουν και μοχλό καινοτομίες και γι' αυτό ακριβώς οι διατάξεις λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίζουν και την καινοτομία. Συμφωνώ επίσης ε, με αυτό το οποίο προτείνουν αρκετοί συνάδελφοι δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τις διατάξεις ε, προϊόντων ε, προστασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης για να έχουμε και για μη γεωργικά προϊόντα μια προστασία βάσει γεωγραφικής ένδειξης. Ε, είμαι λίγο όμως πιο επιφυλακτική για την τροπολογία 28, η οποία ζητά πλήρη εναρμόνιση. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες μεταξύ γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων που σημαίνει ότι θα πρέπει να εμπνευστούμε ε, μεν από τα γεωργικά προϊόντα για να δημιουργήσουμε κάτι αντίστοιχο για τα μη γεωργικά προϊόντα, αλλά δεν θα πρέπει να είναι όλα ταυτόσιμα. Επίσης υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που αναφέρονται στη νέα διαδικασία μελετών, διαβούλευσης κλπ. Εγώ θεωρώ ότι πέρασε ο καιρός των διαβουλεύσεων και των μελετών. Υπήρχε μια πολύ καλή μελάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013 που ήταν πληρέστατη. Ε, και αναφερόταν στην ανάγκη να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες γεωγραφικές ε, ε, ενδείξεις για τα χειροποίητα προϊόντα, καθώς επίσης και κάποια αποτελέσματα τα οποία δημοσιεύτηκαν πριν από ένα μήνα Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη βάση γνώσεων και όπως ε, υπενθυμίζουν και αρκετοί συνάδελφοι στις συμβαστικές ε, τροπολογίες θα προσπαθήσω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσει πλέον στην νομοθεσία και να προτείνει στην καλύτερη δυνατή προθεσμία ένα νομοθετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την επέκταση αυτών των γεωγραφικών ενδείξεων ε, προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν συμβαστικές προτάσεις, ε, τις οποίες όμως θα πλαισιώσω βάσει αρκετών ε, τροπολογιών των συναδέλφων, τις οποίες θα ήθελα να υποστηρίξω. Επίσης θα ήθελα να πω ότι ως προς το νομικό πλαίσιο θα λάβουμε υπόψη μας και τη γνωμοδότηση των συναδέλφων της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, την ανάγκη να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο για να προστατεύσουμε καλύτερα τις γεωγραφικέ ενδείξεις στα πλαίσια των συζητήσεων για τις εμπορικές ε, συμφωνίες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο και επίσης ε, περιμένουμε και τη γνωμοδότηση λοιπόν των συναδέλφων από την Επιτροπή Ίντα αλλά και των Επιτροπών ε, Πολιτισμού και Εσωτερικής Αγοράς που θα έχουν να προσθεθούν λοιπόν στις τροπολογίες που υπευλήθησαν. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις πολύ επικοδομητικές προτάσεις τους και φυσικά δεσμεύομαι να παρουσιάσω τροπολογίες ε, με το μεγαλύτερο δυνατό συμβασμό για τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ο κύριος Μπούντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς ε, να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της αυτή και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να καταφέρουμε να έχουμε νομοθεσία στον τομέα αυτό. Πριν από λίγο λέγαμε πόσο σημαντικό είναι να αισθανόμαστε ότι ανήκουμε πραγματικά σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μία ενοποιημένη Ευρώπη. Από την άλλη όμως θα πρέπει να προασπίσουμε και τη διαφορετικότητα των κρατών μελών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με μία τέτοια έκθεση πετυχαίνουμε αυτή την ευκταία ισορροπία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ξεχωριστή νομοθεσία ξεχωριστή από αυτή που ισχύει για, τα, για τις γεωγραφικές ενδείξεις των γεωργικών προϊόντων. Εδώ αναφερόμαστε σε μη γεωργικά προϊόντα. Θεωρώ και εγώ ότι η νομοθεσία αυτή θα μας επιτρέψει να προασπίσουμε τις αξίες κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε έχει το λόγο. Και εγώ είμαι υπέρα του κειμένου αυτού. Υποβλήθησαν πολλές τροπολογίες οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες και μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε το κείμενο. Νομίζω ότι πραγματικά τονίζουμε εδώ πέρα ήδη από την αρχική εκδοχή του κειμένου το πόσο σημαντικό είναι μέσω του κειμένου αυτού να προασπίσουμε τους καταναλωτές, να καταπολεμήσουμε την απάτη και τις απομιμήσεις, να καταφέρουμε να προωθήσουμε ακόμα και τον τουριστικό τομέα, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον κύκλο εργασιών ορισμένων επιχειρήσεων, πώς μπορούμε επίσης να προασπίσουμε ορισμένες μικρές επιχειρήσεις από τον αθέμητο διεθνή ανταγωνισμό. Ορισμένες τροπολογίες έχουν ως στόχο να διατηρήσουν την εθνική προστασία. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει όντως να διατηρηθεί εφόσον αποτελεσματική, καλή εναρμόνιση, αλλά θα πρέπει να αποτελεί ομοιομορφία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο με τις τροπολογίες 17 και 45 προσπαθώ να εξασφαλίσω αυτό το πράγμα. Ο ορισμός τώρα αυτών των γεωγραφικών ενδείξεων για τα μη γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να είναι ορισμοί σαφείς και συγκεκριμένη, η αρχική εκδοχή του κειμένου που αναφερόταν σε έναν πιο επεκτετικό ορισμό νομίζω ότι θα πρέπει να διορθωθεί με τις συμβαστικές τροπολογίες. Διατρέχουμε και κάποιο κίνδυνο και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε εδώ πέρα προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει αυτή η νέα προστασία να επεκταθεί σε σήματα τα οποία δεν περιέχουν κείμενο, δεν περιέχουν γράμματα, δεν περιέχουν λέξεις, Ας μην πηγαίνουμε πάρα πολύ μακριά και ας είμαστε κυρίως προσεκτικοί. Ας προσέξουμε επίσης λίγο την ε, προστασία που θα δώσουμε για μη γεωργικά ονόματα, για μη τοπονύμια. Εδώ πέρα η τροπολογία 38, την οποία επέβαλα μας καλεί να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και συμφωνώ με την κυρία Ροζιέρ ότι η σφαιρική ολική εναρμόνιση όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα γεωργικά προϊόντα δεν μπορεί εδώ πέρα να εφαρμοστεί κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί φοβάμαι ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε κατά ενό συστήματος το οποίο λειτουργεί μέχρι στιγμής καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Άντερσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι τα συστήματα τα οποία υφίστανται θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε προσεκτικά σε σχέση με τις λεπτομέρειες. Να προσέξουμε να μην γίνουν το κύριο πρόβλημα οι λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο κάπως μας ανησυχεί και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο θέμα του να γνωρίζουμε αν οι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων και εκείνων που δεν είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αν λαμβάνονται δηλαδή υπόψη τα θέματα των γεωργικών προϊόντων και εκείνων που δεν είναι γεωργικά προϊόντα σε σχέση με την αγορά που είναι ελεύθερη και δίνει, ε, παρέχει καλά προϊόντα καλής ποιότητας για τους καταναλωτές. Δεν γνωρίζω αν αυτό μπορεί να επεκταθεί και στον μη γεωργικό προϊόν, ε, στα μη γεωργικά προϊόντα. Αν θα μπορούσε δηλαδή να διασφαλιστεί και η ποιότητα και ο ανταγωνισμός. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην υπερβολικά περιοριζόμαστε μέσα στο πλαίσιο αποκλειστικά των γεωργικών προϊόντων. Αυτό είναι μία, η μία πλευρά που θα ήθελα να αναφέρω. Από την άλλη πλευρά, ίσως είναι νωρίς να πει κανείς ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο τέλος ή όχι. Ευχαριστώ. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο. Δεν βλέπω να ζητούν άλλοι τον λόγο. Η κυρία Ροζιέρ παρακαλώ θα ήθελε να ολοκληρώσει ο κύριος Δεγκράντες παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Ζητώ και συγγνώμη γιατί ε, βιάστηκα να έρθω και ίσως καθυστέρησα λίγο. Εκπροσωπώ σε αυτή την περίπτωση ε, τον συνάδελφο Στάς που δεν ε, μπόρεσε να παραστεί και που με παρακάλεσε να παρέμβω και έχει ανηλυμένες ε, υποχρεώσεις δεν μπορεί να παραστεί και έτσι θα εκθέσω λοιπόν τις θέσεις αυτές. Είναι λοιπόν θετική η ε, προσέγγιση αυτή και δεν είναι το θέμα του να πει κανείς ότι έχουν αλλάξει τα κριτήρια. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε εκείνο το οποίο ξεκίνησε ε, προηγούμενα. Και οι τροπολογίες του ΕΛΚΑ και από πλευράς σας κοιόδους εισηγητού οι προσωπικές ας το πω εσύ συνεισφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής είναι το κριτήριο το οποίο έχει υιοθετηθεί από πλευράς του ΕΛΚΑ σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αναφέρομαι στις τροπολογίες αυτές που είναι συμπληρωματικές θα έλεγα και που προσπαθούν να βελτιώσουν το πλαίσιο, το περιεχόμενο της κυρίας εισηγήτριας. Και γι' αυτό απλά θα περιοριστώ μια και δεν είναι δική μου η παρέμβαση αυτή, αλλά εξ ονόματος του συναδέλφου, στην αναφορά των κριτηρίων όσον αφορά τα, την προσέγγιση για τις ε, τροπολογίες ε, που έχουν κατατεθεί και τις, ε, τις τροπολογίες συναδέλφου. Τηλεγραφικά θα αναφερθώ στα θέματα αυτά για να μην μακρηγορήσω. Πρώτον, πρόθεση του συναδέλφου είναι να υπάρξει αυτή η προστασία για τα γεωργικά προϊόντα που ρυθμίζονται ήδη στο πλαίσιο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μετατεθεί αυτό το πλαίσιο το προστατευτικό και στα μη γεωργικά προϊόντα. Θετικό είναι αυτό ο στόχος, θα πρέπει λοιπόν να, να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό για να λειτουργήσει σωστά. Επίσης στις τροπολογίες θα πρέπει να εξειδικεύσουμε κάτι το οποίο είναι προφανές αλλά που είναι αναγκαίο να το αναφέρουμε για την ε, παραγωγή και αναγνώριση των προϊόντων αυτών από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δημιουργεί πρόσθετη αξία και γι' αυτό αξίζει τον κόπο να δούμε αυτά τα ποιοτικά προϊόντα και να δούμε και σε σχέση με τις επιμέρους περιοχές παραγωγής αυτών των προϊόντων υπό τους όρους που προτείνει η συγκήτρια αλλά και υπό τους όρους των τροπολογιών που προτείνονται. Επίσης ε, η ε, φήμη μιας τέτοιας γεωγραφικής ένδειξης είναι και μια συλλογική αξία που έχει ένα, μια συλλογική βάση και δημιουργεί ένα κύρος και έχει προταχικό χαρακτήρα αυτό για τους καταναλωτές. Επίσης, σε σχέση με τις τροπολογίες, οι γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να έχουν και ένα δυναμικό οικονομικό και πρέπει να το δούμε και αυτό. Δεν είναι ίσονος σημασία αυτό. Στο τέλος τέλος εργαζόμαστε επιθεμάτων που μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι τόσο ουσιώδη και όμως έχουν τη σπουδαιότητά τους. Μπορούν να δημιουργήσουν ε, ωφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν να δούμε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν αυτές οι προτάσεις σε αυτό το πλαίσιο και με τη δημιουργία μιας γεωγραφικής ένδειξης που πρέπει να ε, είναι ε, θέμα το οποίο θα χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές και να μπορέσουμε να ζητήσουμε να ε, στρέψουμε την προσοχή μας σε θέματα προαγωγής αυτών των προϊόντων. Στο τέλος θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στο να υπάρξει και ένα καθεστώς ε, εποπτείας για τις παραβάσεις και παραβιάσεις και κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται. Δεν είναι δυνατόν να είναι αποτελεσματικό το πλαίσιο προστασίας αν δεν ε, υπάρχει αποτελεσματική εποπτεία με κυρώσεις. Ε, αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη σε σχέση με την πραγματικότητα. Δεν πρέπει λοιπόν να μελήσουμε αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Και πιστεύω ότι σε σχέση με την ε, κυρία εισηγήτρια, στρέφομαι σε εσά κυρία εισηγήτρια, διότι εσείς είσαστε τελικά η υπεύθυνη, αρμόδια που θα επιλέξει τα κριτήρια για τις προτάσεις που κατατίθενται από τον έναν ή άλλον. Και σε σχέση με την ε, σκιώδη εισήγηση από πλευράς, του, από συναδέφου είναι όλες ε, επικοδομητικές αυτές οι τροπολογίες και νομίζω ότι μπορούν ε, να αξίζουν να ενταχθούν σε συμβαστικές τροπολογίες οι προτάσεις αυτές ώστε να τύχουν ευρύτερης έγκρισης, ευρύτερης συνένεσης. Βασίζομαι λοιπόν στις ικανότητες της εισηγήτριας για να μπορέσει να εμπλουτιστεί η έκθεση με αυτά τα κοινά στοιχεία της κοινή αυτής ε, ε, προαίρεσης και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο να διασφαλίσουμε την ε, κληρονομιά μας σε σχέση με αυτά τα προϊόντα. Και θα συνεισφέρει αυτό και για την απασχόληση με σημαντικό τρόπο. Είναι στο χέρι μας να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Έχουμε κάθε εμπιστοσύνη στην εισηγήτρια να μπορέσει, ότι θα μπορέσει να συνενώσει τα στοιχεία αυτά με βάση τις προτάσεις του ενός ή του άλλου και να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Και έτσι λοιπόν θα εμπλουτιστεί η έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία θέλει να πάρει το λόγο και πάλι. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις εξηγήσει που έκαναν για τις τροπολογίες τους και να πω ότι πραγματικά θα προσπαθήσω να έχω με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία λοιπόν. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα για σήμερα το απόγευμα και μπορούμε να συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών, η οποία θα γίνει και κλεισμένα των θυρών. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, συμμετοχή σας.